Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. like first to welcome Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο εμπειρογνώμονες που θα πάρουν το λόγο σήμερα. Τον κύριο Γκέργεφ, τον κύριο Ανιέλη και τον κύριο Καπόνε. Θα σας τους παρουσιάσουμε τον καθένα από αυτούς πριν από την ομιλία τους. Η ακρόαση αυτή έχει σχέση με τα σημαντικά θέματα ε, με το λεγόμενο 5G, κινητή τηλεφωνία πέμπτου επίπεδου, πέμπτης γενεάς, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, νέες τεχνολογίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια νέα υπηρεσία που βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Να ευχαριστήσω τα μέλη της ΣΥΤΡΕ, τα οποία ασχολήθηκαν με τα θέματα της 5G, με διαφορετικούς κανονισμούς τα τελευταία χρόνια. Την κυρία Πιλάρτε Καστίγιο Βέρα, τον κύριο Μπόνι, την κυρία Κουμπούλα Νάτρη, να σας ενημερώσω επίσης ότι έχουμε δυόμιση ώρες στη διάθεσή μας για την συγκεκριμένη ακρόση. Θα ήθελα οι εμπειρογνώμονες να μην ξεπεράσουν τα 10 λεπτά ο καθένας και τα μέλη επίσης θα πρέπει όταν πάρουν το λόγο να περιορίσουν και αυτά το χρόνο τους για να μπορέσουν οι ομιλητές να δώσουν τις απαντήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σορίνιο ως εισηγητής. Έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του ο κύριος Σορίνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω και τους συμμετέχοντες στο πάνελ αυτής της ακρόσης. Ο τίτλος είναι «Συνδεσιμότητα του ψηφιακού μέλλοντος». η, το ψηφιακό μέλλον θα πρέπει να συνοδεύεται από, μια, από ένα συγκεκριμένο πολιτικό όραμα και σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουμε καθυστερήσει. Δεν διαθέτουμε επαρκή προπολογισμό για να καλύψουμε εύκολα τη διαφορά από άλλες επιστημονικές και οικονομικές δυνάμεις. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των ομιλητών συγκεκριμένα για, την, ε, για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ. Το αποτελεί μια απειλή λοιπόν. Αυτή την απειλή όμως θα πρέπει να την μετασχηματίσουμε. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε. Η αντιγραφή δεν είναι λύση. Χρειάζεται να καινοτομήσουμε και να διδαχθούμε από αυτά που έχουμε μάθει άλλοι. Συνδεσιμότητα στο μέλλον σημαίνει διαφάνεια, ε, να εστιάσουμε στους ανθρώπους, στις ανάγκες τους, ε, με υψηλές προδιαγραφές, ηθικές προδιαγραφές και πλήρη πρόσβαση για όλους. Έχουμε δύο σημαντικά προγράμματα, δύο εκθέσεις για την συνδεσιμότητα. Εγώ είμαι η του, του, 5 του G54U. Είναι πολύ σημαντική ε, αυτή η πρωτοβουλία. Το Wi-Fi4U, όχι G54U, Wi-Fi4U. Ε, στόχος μας είναι υψηλή ποιότητα υπηρεσίες ε, με ευρία πρόσβαση σε αυτές και μια ψηφιακή ευρωπαϊκή ταυτότητα ισχυρή. Νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και την καθυστέρηση. Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, τέλος, έχουμε το πρώτο πρόγραμμα το οποίο έκλεισε στον τριμερή διάλογο για τον νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 με τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν η, Ευρωπα... η ψηφιακή Ευρώπη. Ήμουν σκιώδης ηγητής σε αυτό το πρόγραμμα και το γεγονό ότι καταφέραμε και το διαπραγματευτήκαμε ένα φιλόδοξο ε, πρόγραμμα για το μέλλον της Ευρώπης και είναι σημαντικό για την επόμενη δεκαετία και αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολιτική βούληση άρα λοιπόν και οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει στην ψηφιακή εποχή και να συνδέσει το μέλλον της με τους πολίτες της. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο διαφορετικά τμήματα θα ακολουθήσουν. Πριν γίνει αυτό όμως, θα δώσω το λόγο στην κυρία Πιλάρντε Καστίγιο Βέρα, εισηγήτρια για τα θέματα των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη. Χωρίς μικρόφωνο η κυρία Καστίγιο Βέρα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Τα θέματα της συνδεσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε η Ευρώπη να ηγηθεί της κοινωνίας των gigabit. Είναι πολλά τα παραδείγματα των τομέων ε, που έχουν, ε, ε, στους οποίους θα έχει υψηλή ζήτηση η ασφαλής και γρήγορη συνδεσιμότητα. Με το παρόν στάτους κβο η Ευρώπη δεν θα είναι δυστυχώς σε θέση να ανταποκριθεί στις δομές οι οποίες απαιτούνται. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 500 με 600 δις, τα 90% φυσικά θα διατεθούν από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η ε, ευκαιρία αυτή. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, να ελέγξουμε δηλαδή όλες τις δυνατότητες, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, να δημιουργήσουμε δίκτυα υψηλής αξιοπιστίας και να διαμορφώσουμε ένα διακανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα θέσει τις προϋποθέσεις για σωστές νομοθετικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει το νέο πλαίσιο να δίνει την δυνατότητα στην αγορά να επιλύει τα προβλήματα, να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες και να βοηθά να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στις εταιρείες που διαχειρίζονται την, τις νέες αυτές επικοινωνίες. Έτσι ταυτόχρονα θα πρέπει να διαθέσουμε ελεύθερα φάσματα πεδίου έτσι ώστε να επιτρέψουμε στα κινητά δίκτυα 5G από 3,3 μέχρι 26 GHz πριν το 2030. Στην Ευρώπη λοιπόν βρισκόμαστε σε μια ειδική κατάσταση να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση ε, πρώτης τάξεως θα έλεγα. Έχουμε μία αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, έχουμε ένα ΑΕΠ ακόμα και σήμερα το οποίο αντιπροσωπεύει 20 23% του παγκόσμιου ΑΕΠ και έχουμε και μια ανταγωνιστική βιομηχανία παγκοσμίως Έχουμε δηλαδή ε, την ευκαιρία να προχωρήσουμε και η συνδεσιμότητα είναι προϋπόθεση θα έλεγα για να μπορέσουμε να περάσουμε στην πλήρη ψηφιοποίηση της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ κυρία Ντελκαστίγιο. Πράγματι είπατε ότι ε, ε, είναι η πρώτη φορά που έχουμε την δυνατότητα αυτή ε, που θα είμαστε πρωτοπόροι στον κόσμο. Εγώ πέρασα όλη μου τη ζωή στη, στα ηλεκτρονικά και μακάρι να το πετύχουμε. Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα δώσω το λόγο στους δύο πρώτους ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο Αντώνιο Καπόνε. Είναι καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Μιλάνου. Θα μας κάνει μια παρουσίαση της 5G και θα μας παρουσιάσει τις διαφορές ανάμεσα στις ε, υπάρχουσες γενναίες δικτύων και στις μελλοντικές γενναίες δικτύων. Κύριε Καπόνε, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τιμή μου που με καλέσατε. Τα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να απαντήσω μερικά από τα βασικά ερωτήματα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι σχετικά με το 5G, με την τεχνολογία 5G. Ας ξεκινήσω λοιπόν από μια γενική ερώτηση. Γιατί η τεχνολογία αυτή είναι διαφορετική από τις προηγούμενες γενιές. Κατά την άποψή μου, τρεις είναι οι διαφορές. Αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ είναι το τρίγωνο της πέμπτης γενιάς του 5G. Είναι ένας τρόπος να περιγράψουμε την πέμπτη γενιά τη χρησιμοποιούμε για να δείξουμε πόσες διαφορετικές εφαρμογές μπορούμε να υλοποιήσουμε. Ε, είναι όμως τρίγωνο, δεν είναι τετράγωνο ούτε κύκλος και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ο βασικός λόγος είναι ότι η πέμπτη γενιά για πρώτη φορά δεν βελτιώνει μόνο τις ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων, αλλά και άλλες διαστάσεις. Για παράδειγμα, ε, αξιοπιστία και καθυστέρηση και από την άλλη μεριά έχουμε τον αριθμό των χρηστών και, των, ε, και την ε, κατανάλωση ενέργειας. Οπότε η πρώτη διαφορά που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η πέμπτη γενιά μπορεί να διαχειρίζεται πολλές διαφορετικές συνθήκες εργασίας και να εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό εφαρμογών πρωτοφανές στην ιστορία. Πρωτοφανή στην ιστορία. Δεύτερη πτυχή που πρέπει να ε, σχολιάσω είναι ότι χρησιμοποιεί τεχνολογίες ε, δημιουργίας εικονικών ε, δικτύων και πάνω στην ίδια υποδομή μπορεί να δημιουργήσει ένα αριθμό, μεγάλο αριθμό ε, εικονικών δικτύων τα οποία το καθένα θα έχει διαφορετικές ανάγκες και θα εξυπηρετείται από διαφορετικές εφαρμογές. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές ε, ε λειτουργίες εξυπηρέτησης ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Δεύτερη λοιπόν διαφορά είναι ότι με την πέμπτη γενιά έχουμε ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να κατατμηθεί σε φλίδες, αν θέλετε να το δούμε έτσι, σε φέτες εικονικών δικτύων τα οποία μπορούμε, μπορούν να τα διαχειρίζονται νέοι πάροχοι. Η πέμπτη γενιά θα κάνει πλήρη χρήση του edge computing, δηλαδή ε, ικανότητα διαχείρισης δεδομένων πολύ κοντά στο χρήστη. Η διαφορά είναι λοιπόν ότι η πέμπτη έννοια δεν δίνει απλώς κανάλια για, τη, για την ε, διακίνηση δεδομένων, αλλά πλατφόρμες πάνω στις οποίες θα τρέχουν εφαρμογές που θα, και θα παρέχονται υπηρεσίες. Δηλαδή το δίκτυο γίνεται πλέον μια προγραμματιζόμενη πλατφόρμα ε, που θα είναι ε, διαθέσιμη για εφαρμογές προς το χρήστη, που θα προσφέρονται στο χρήστη. Αυτή είναι η βασική λόγη για τους οποίους οποίους η πέμπτη γενιά δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες. Το ερώτημα είναι όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό, κρίσιμο για την ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία το να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει η πέμπτη γενιά. Έχουμε, μιλάμε για την ψηφιακή το ψηφιακό μετασχηματισμό εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η προχωρημένη συνδεσιμότητα που δίνει η πέμπτη γενιά είναι το στοιχείο κλειδί το οποίο έλειπε μέχρι τώρα. Μπορεί αυτό τόσο καινούριο κρίκο να αλλάξει τελείω το πανόραμα, το τοπίο. Ο τεράστιο αριθμό ε, εφαρμογών που σχεδιάζονται ή μπορούν να σχεδιαστούν στο πλαίσιο του 5ης γενιάς θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό κλάδων της οικονομίας. Επιπλέον, μπορούμε να πούμε ότι η πέμπτη γενιά μπορεί να δώσει το θα που χρειάζεται το μυαλό της τεχνητής νοημοσύνης. Αν δεν έχουμε τα μέσα για να εφαρμόσουμε τα δεδομένα της, της ε, νοημοσύνης δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε οι ευκαιρίες αυτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η διαθεσιμότητα, της, ε, ε, η διαθεσιμότητα δικτύων σε παντού μειώνει τα εμπόδια που υπάρχουν στην εισαγωγή καινούριων καινοτόμων λύσεων. Ας σκεφτούμε startups, μικρές καινούριες ε, εταιρείε στην Ευρώπη, ε, οι οποίες θα ωφεληθούν πάρα πολύ όταν υπάρχει ένα δίκτυο που θα προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες ήδη. Άρα λοιπόν οι ιδέες τους θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν. Όπως τα smartphones έδωσαν μια πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίστηκε μια ολόκληρη οικονομία εφαρμογών, έτσι και η πέμπτη γενιά μπορεί να δώσει να αποτελέσει την πλατφόρμα ε, για ψηφιακές εφαρμογές στο φυσικό κόσμο. Αντίθετα με το παραδοσιακό ίντερνετ, που ωφελούσε τους μεγάλους ε, παγκόσμιους παίκτες, ε, η πέμπτη γενιά θα είναι πιο τοπική, γιατί συνδέεται πολύ περισσότερο με το φυσικό κόσμο και με τις εφαρμογές οι οποίες θα έχουν σχεδιαστεί για, το, για την πέμπτη γενιά. Θα, αυτές οι ε, εφαρμογές θα εξυπηρετούν την παγκόσμια αγορά, αλλά και την τοπική αγορά. Γι' αυτό το λόγο θα δημιουργηθούν και θα προγραμματιστούμε πάνω σε τοπικά οικονομικά οικοσυστήματα. Άρα λοιπόν η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ευκαιρία να διατηρήσει την προσθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί από την πέμπτη γενιά και να μην την αφήσει να πετάξει για άλλες επικράτειες. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει και κάποιες δοκιμές της πέμπτης γενιάς. Οπότε η τέταρτη ερώτηση είναι ποια είναι τα διδάγματα τα οποία πήραμε από αυτές τις δοκιμές στην Ευρώπη. Ε, εγώ συμμετέχω σε μια δοκιμή που γίνεται στη Μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνου. Ε, η δοκιμή αυτή γίνεται από τη Vodafone με 28 εταίρους και 10 δημόσιους οργανισμούς με επένδυση συνολικά πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά για τη δοκιμή. Έχουμε 41 ε, περιπτώσεις διαφορετικών χρηστών ε, σε 7 τομείς. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς δημιουργούνται καινούργιε λύσεις και αλλάζει ο ρόλος ε, των παρόχων. οι δοκιμές αυτές επιτρέπουν την έκφραση καινούριων ιδεών, διότι ακριβώ δημιουργούμε ήδη μια υποδομή πάνω στην οποία αυτέ οι ιδέε μπορούν να υλοποιηθούν. Η ερώτηση είναι βέβαια, μπορούμε με αυτέ τι δοκιμέ να εντοπίσουμε αν υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη τη πέμπτη γενιά. Ειλικρινά να σα πω ότι τα ωφέλη αυτή τη καινούρια υποδομή που δίνει η πέμπτη γενιά δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά επί και το να χτίσει κανείς μια εφαρμογή δεν είναι απλό πράγμα. Απ' την άλλη μεριά είναι ακόμα πιο δύσκολο αν όταν κανείς θέλει αυτές οι ιδέες να τις κάνει και επιχειρηματικά μοντέλα, βιώσιμα. Οπότε θα αλλάξουν οι σχέσεις ανάμεσα στην, ε, στη στην τηλεπικοινωνική βιομηχανία και τους άλλους κλάδους οικονομίας. Θα πρέπει να βασιστούμε στο ανοιχτό μοντέλο καινοτομία, το οποίο θα πυροδοτήσει την καινοτομία σε αυτό το τομέα. Τελευταία ερώτηση. Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Στις περισσότερες χώρες η πέμπτη γενιά θα μπει στο εμπόριο, θα βγει στην αγορά. Μετά από κάποια χρόνια ερευνών πια, σύντομα θα φτάσουμε στην δυνατότητα εμπορικοποίησης ε, αυτής της τεχνολογίας. Αυτή είναι μια κορυφή. Ε, μετά η αλλά αν νομίζουμε ότι αυτό είναι το τέλος της διαδρομής και ότι οι επιχειρήσεις θα πάρουν την σκητάλη και θα την εξελίξουν, είναι λάθος. Τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για να αντιληφθούμε το πόσο από το δυναμικό αυτής της τεχνολογίας μπορεί να μεταφραστεί στην πραγματική οικονομία. Και εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του κράτους και των πολιτικών του των κρατικών πολιτικών. Μία από τις βασικές προκλήσεις που έχουμε είναι η προώθηση των επενδύσεων. Γιατί, γιατί χρειάζεται τα δίκτυα να αναπτυχθούν γρήγορα. Άλλο το δίκτυο να είναι έτοιμο σε τρία χρόνια και άλλο σε δέκα. Όπως γνωρίζετε η ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών δικτύου είναι ένα, μία από τις πιο ανταγωνιστικές του κόσμου. Αυτό είναι ωφέλιμο βέβαια για τους τελικούς χρήστες, αλλά όχι απαραίτητα για τους επενδυτές, ιδιαίτερα αν δεν την διαχειριστούν σωστά. Έχουμε και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, σχετικό ιδιαίτερα με τη χώρα μου, έχουμε διαφορετικά όρια σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Αυτό μπορεί να είναι θέμα. Γιατί οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ε, μπορούν να κοστίσουν πάρα πολύ, νόμοι δηλαδή για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές μπορούν να κοστίσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη του δικτύου. Η συνεργασία είναι κλειδί. Το να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και άλλους τομείς οικονομίας θα αποδειχθεί κρίσιμο στο μέλλον. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε επίσης τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων. Και οι διαφορές στις τοπικές οικονομίες και τις τοπικές κουλτούρες στην Ευρώπη μπορούν να δώσουν λύσεις σε αυτή την καινούργια ψηφιακή οικονομία, οι λύσεις οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε την συνεργασία και τη δημιουργία και την, συγγνώμη, και τη χρηματοδότηση που χρειαζόμαστε ε, για καινούριε επενδύσεις. Χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν εταιρείε startup, διότι γνωρίζετε ότι σε αυτό το θέμα υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω συμπέρασμα, να σα συνοψίσω τα εξή. Η πέμπτη γενιά είναι πραγματικά μια ευκαιρία για την Ευρώπη για να ανακτήσει ένα δεσπόζοντα ρόλο στην ψηφιακή οικονομία οι ευρωπαϊκές διαφορές ε, που έχουμε σε τοπικό επίπεδο ε, σε ό,τι αφορά την πέμπτη γενιά μπορούν να ε, γίνουν πλεονέκτημα αν τις διαχειριστούμε σωστά. Οι κρατικές και δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα γίνουν επαρκείς επενδύσεις σε υποδομές και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει μικρόφωνο ο πρόεδρος, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Η πιο σημαντική φράση που είπατε ήταν αν θα εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η πέμπτη γενεά της ε, διασύνθεσης των... Νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ομιλητή, να δώσω τον λόγο στον κύριο Γεωργίευ, Public Policy Manager του GMSF, που θα εξηγήσει τα ωφέλη και εμπόδια μελλοντικών δικτύων 5G. Κύριε Γεωργίευ, σας δίνω 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Είναι πραγματική χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα για να μπορέσω να εξηγήσω το σημαντικό αυτό θέμα. Η GSMA βάλει πολλές εκατοντάδες operators όλο τον χρόνο και 250 εταιρείε που συμμετέχουν στα ευρεία δίκτυα. Και κάτι που κάνουμε είναι ότι βοηθούμε τις κυβερνήσεις για να μπορέσουν να διασυνδέσουν τους πάντες και τα πάντα προς την κατεύθυνση ενός μέλλοντος. Να μου επιτρέψετε να αρχίσω την παρουσίαση δείχνοντας ποιοι είναι οι στόχοι του κλάδου για την εποχή των 5G. Δηλαδή θα θέλαμε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ανεφόρον διασυνδεσιμότητα, να υποστηρίξουμε ένα πλήθος δραστηριοτήτων στην κοινωνία, να δώσουμε νέα δίκτυα με οικονομικό τρόπο, είτε ανεξάρτητα είτε μέσα σε κοινοπραξίες, να επιταχύνουμε την μετατροπή των ε, βιομηχανιών, των κάθετων βιομηχανιών, προωθώντας την ψηφιοποίηση και αυτοματισμούς, να φέρουμε μια πραγματική επανάσταση στην εμπειρία του κινητού ευρέως φάσματος, με νέες υπηρεσίες και τέλος να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν νέες χρήσεις για παράδειγμα για FEIUT μέσα σε πλήθος σενάριο και να προσφέρουμε μια πλατφόρμα για τις ε, κρίσιμες ε, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Έχοντας υπόψη το όραμα αυτό, αυτό που κάναμε πέρσι ήταν μια έρευνα όπου ζητήσαμε από τους καταναλωτές 16 ε, χωρών ανά τον κόσμο τι αναμένουν από το 5G και βλέπετε στον ε, πίνακα αυτό, στο γράφημα αυτό, είχαν δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικές ε, ε, απαντήσεις και βλέπουμε ότι παραπάνω από τους μισούς αναμένουν υψηλότερες ταχύτητες και καλύτερη κάλυψη. Θα ήθελα όμως να έρθω τώρα λίγο πού βρίσκεται η Ευρώπη τώρα. Γιατί έχουμε και την intelligence μονάδα μας η οποία εξετάζει τις προβολές των 5G για όλο τον κόσμο μέχρι το 2025 και αυτό που σας δείχνω στην διαφάνεια είναι, ενώ θα ηγείται η Νότια Κορέα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, όπου περιμένουμε οι διασυνδέσεις 5G να είναι της τάξης του 60%, θα ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, Βλέπετε στον πίνακα ότι ο μέσος όρος ε, της Ευρώπης των 28 ε, προηγείται της Κίνας. Αυτό που βλέπετε στην διαφάνεια είναι ότι οι τέσσερις αυτές μεγάλες οικονομίες που περιλαμβάνεται και η Ευρώπη των 28 θα φτάνουν το 70% των διασυνδέσεων 5G μέχρι το 2025. Τώρα μπορεί να αναλυθεί το νούμερο αυτό κάπως καλύτερα και να δείξω την ανισότητα μεταξύ των χωρών μελών εδώ στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενώ πολλέ τα πάνε πάρα πολύ καλά, σε σχέση για παράδειγμα με την Ιαπωνία ή τι Ηνωμένε Πολιτείε, βλέπουμε ωστόσο τα δύο τρίτα περίπου των χωρών μελών που θα βρίσκονται κάτω του μέσου όρου και ένα τρίτο περίπου θα είναι τα μισά του μέσου όρου της Ευρώπης. Ε, θα ήθελα τώρα να έρθω κυρίως στα εξής θέματα πολιτικής δηλαδή και ποιες θα είναι οι προκλήσεις για τις πολιτικές αυτές. Πολύ σύντομα για την εφαρμογή του κώδικα, ορισμένες από τις τεχνικές ε, προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε και θέματα εφαρμογής του κώδικα στην Ευρώπη. Πριν να προχωρήσω τώρα στον κώδικα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε για την πολύ και καλή δουλειά που έχετε κάνει στην προσπάθεια να εξασφαλίσετε ένα γερό θεμέλιο για την εξέλιξη αυτή στην Ευρώπη. Γνωρίζω ότι έχει δοθεί η τελική μορφή και είναι πολύ σημαντικό στην πρόταση και οι χώρες ε, μέλη πάνε να την εφαρμόσουν ε, με πραγματικά τα βλέμματα στραμμένα στο μέλλον. Αφενός τώρα σε ό,τι αφορά τους φιλόδοξους στόχους των χωρών μελών και εμείς αναμένουμε πραγματικά γνήσια ωφέλη του 5G υπέρ των πολιτών και της οικονομίας και του ηγετικού ρόλου και της διάθεσης να θυσιάσουν οι χώρες μέλη βραχυπρόθεσμα κέρδη για να ε, καταλήξουν σε υψηλά μακροπρόθεσμα ωφέλη. Ξεκινώντας το με το φάσμα, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς το εξής. Το φάσμα στην Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει ώστε το 5G να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα ή μπορεί και να το παρεμποδίσει. Το έχουμε αποδείξει αυτό σε τέσσερις τομείς. Σε τέσσερις Αυτό που έχει σημασία για το φάσμα στην Ευρώπη είναι ότι χρειάζεται επαρκές φάσμα, άδειες, αδειοδότηση δηλαδή υπό τους σωστούς όρους και στη σωστή τιμή. Σε ό,τι αφορά την προσφορά, είναι σημαντικό να, υπάρχει, να υπάρχουν επαρκή block ανά operator, ώστε να μπορέσει το 5G να εξασφαλίσει τις ταχύτητες που αναμένουν οι καταναλωτές. Μιλούμε για 80% MHz στην ζώνη C και περίπου 1 GHz στην ζώνη των 26 GHz. Για τους όρους τώρα είναι σημαντικό όταν θα διοδοτηθούν οι συχνότητες αυτές να είναι ρεαλιστικές και δυνατόν να επιτευθούν οι ε, ε, συνθήκες που θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, επιβραβεύσεις. Πριν από λίγες εβδομάδες εκδώσαμε έγγραφο πολιτικής σχετικά με το ποιες θα είναι οι θεμελιώδεις βέλτιες πρακτικές για τις ε, αδειοδοτήσεις και δεν μιλάμε για τις αναθέσεις μάλλον, για τις παραχωρήσεις ακόμα καλύτερα και δεν μιλάμε εδώ για δημοπρασίες. Εφόσον κάποιος ζητήσει για μια παραχώρηση, θα πρέπει αυτό να οδηγεί σε βελτίωση της οικονομίας και της αγοράς. Και τέλος το θέμα, των τιμολογίων. Είδαμε από την έρευνα που έχουμε διεξαγάγει και από άλλες ανεξάρτητες έρευνες τον... τις επιπτώσεις των τιμών και των ετήσιων τελών και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτό που ακούμε εδώ σχετικά με τις τιμές είναι ότι οι τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερη ε, ε, διασυνδεσιμότητα και λιγότερο σε άμεσο έσοδο υπέρ των κυβερνήσεων. Τώρα υπάρχουν και ορισμένα τεχνικά θέματα και προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη για τα 26 GHz που είναι και από τα πιο, πιο, σημαντικές, πιο σημαντικές ζώνες του φάσματος. Η επιλογή των χωρών μελών σε ό,τι αφορά του τεχνικού αυτούς όρου ήταν υπερβολικά συντηρητική και υπερπροστατευτική. Και έχει σημαντική επίπτωση στην ικανότητα του κλάδου να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Όταν μιλούμε για τη ζώνη σε, υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα defragmentation, του, της αναστροφής του κατακαιρματισμού δηλαδή ενώ είχε εναρμονιστεί η ζώνη C σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Όμως διάφοροι χρήστες χρησιμοποίησαν διάφορα τμήματα του φάσματος αυτού. Θα έπρεπε να ε, επέλθει η, αυτό, η defragmentation το δυνατόν συντομότερο. Τέλος, θα χρειαστεί να εξεταστεί και ο συντονισμός και διαμεθοριακός. Αυτό είναι σημαντική πρόκληση, διότι η Ευρώπη νομίζω δεν διαθέτει εμπειρία στην χρήση τέτοιων ζωνών συχνοτήτων και αυτό ενδέχεται να οδηγήσει τον κίνδυνο να μείνουν μεγάλες περιφέρειες χωρίς κάλυψη. Προχωρώ τώρα στις ε, προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ανάπτυξη και θα σας παρουσιάσω δύο διαφορετικά θέματα. Κάτι που ακούσατε και πριν, που είναι η πολιτική ΕΜΕΦ e εξετάστε και τον σχετικό πίνακα, βλέπετε τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζονται στις, ε, στα διεθνή πρότυπα του 1999 και ως αποτέλεσμα αυτό που έχουμε είναι ένα τρίτο περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσμού να θίγεται, να πλήττεται μάλλον από λιγότερο αποτελεσματικά δίκτυα και εάν δεν διορθωθεί θα παρεμποδίσει και την εφαρμογή του δικτύου 5G. Το δεύτερο που είναι σημαντικό έχει σχέση με την sighting policy. Αυτό που βλέπουμε εδώ, εξετάσαμε δηλαδή διαφορετικές χώρες μέλη και τις πολιτικές τους και σε ό,τι αφορά πόσο χρειάζεται για να αδειοδοτηθεί η λειτουργία μιας, ενός, ενός βασικού σταθμού base station. Και θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ποικίλα, ποικίλες διαστρωματώσεις εθνικών αρχών, κεντρικών και περιφερειακών, που οδηγεί τελικώ σε μια βαριά γραφειοκρατία που καθιστά δύσκολη την ταχεία ανάπτυξη του δικτύου 5G. Με, πρόκειται για συντηρητική πρόβλεψη εδώ, αλλά όταν μιλούμε για 5G θα πρέπει τα sites να αυξηθούν σημαντικά και μιλώ εδώ για δύο τρεις φορές. Η FCC όμως Επιτροπή μιλά συχνά για 200 φορές περισσότερο και ταχύτερα. Αν αυτές οι πολιτικές λοιπόν δεν εναρμονιστούν και απλουστευτούν θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν. Το άρθρο 57 του κώδικα για μικρέ κυψέλε είναι πάρα πολύ σημαντικό και με κανένα τρόπο δεν είναι όμω η πανάκια που θα επιτρέψει να εντατικοποιηθούν τα, τα δίκτυα. Αυτό που χρειάζεται ακόμα είναι η δυνατότητα όχι μόνο για μια αναβάθμιση αλλά να υπάρχουν και οι mm. λεγόμενες microsites για τον απλό λόγο ότι αυτό θα επιτρέψει στους ε, operator κινητών να χρησιμοποιήσουν όλε τι διαθέσιμε συχνότητε 700, 800, 900, 1800 και ούτω καθεξής που σημαίνει ότι θα υπάρχουν πρόσθετα στρώματα κάλυψης. Θα ήθελα τώρα να καταλήξω και μια κάπως θετική νότα, λέγοντας ότι τελικώς όλες αυτές οι προκλήσεις αποτελούν και ευκαιρίες, διότι είναι στα χέρια των χωρών μελών και της ικανότητάς τους να εξετάσουν προκλήσεις αυτές συλλογικά και να παίξουν ένα φιλόδοξο πρωτοπόρο ρόλο. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία για την ώρα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική συντροφικότητα. Δηλαδή χρειαζόμαστε πραγματική αλληλεγγύη και ηγεσία σε στήριξη των ΜΕΝΑ από τους δε και όχι απλώς να συνεργαζόμαστε αλλά κυρίως να εξετάζουμε το τι συμφέρει την χώρα μας. Θα πρέπει λοιπόν σε συλλογική, μέσα από συλλογική προσπάθεια να κάνει το επόμενο βήμα η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Δύο θέματα δεν με εκπλήσουν. Καταρχάς το ότι η Γερμανία είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν το ήξερα αυτό. Αν ακούτε τους Γερμανούς πολιτικούς πιστεύετε ότι είμαστε πρωτοπόροι και απ' την άλλη μόνο το 22% ε, αναμένουν μείωση του κόστους και αυτό με εκπλήσει. Καλώς έχουμε την δυνατότητα τώρα να θέσουμε ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες. Η κυρία Ντελκαστήγιο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές. Αναπτύξατε διαφορετικά θέματα από διαφορετικές πλευρές, μας δώσατε μια πλήρη εικόνα. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση στον κύριο Καπούτο και η άλλη για τον Γκέργκεφ. Προσπαθώντας να ορίσει κανείς να σχεδιάσει το νέο τοπίο του 5G, και στα πλαίσια των εξηγήσεων που δίνεται για, την κρίσιμη, για τον κρίσιμο ρόλο που παίζει αυτή η νέα εικόνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είναι συχνό σήμερα να συναντάτε ένα κάποιο σκεπτικισμό στον τομέα των επενδύσεων. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές επιχειρήσεις και μεταφορές δεδομένων και τηλεπικοινωνιών ε, που δέχονται, που παραδέχονται μάλλον ότι οι επενδύσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε είναι ιδιαίτερα υψηλές και δεν είναι κάτι το οποίο είναι συμβατό με την επιχειρηματικότητα που μας διακρίνει. Συναντάτε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις το διαδίκτυο των πραγμάτων σαν παράδειγμα είναι κάτι το οποίο είναι ελκυστικό για τις εταιρείε αυτές. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη και γι' αυτό διαρωτώμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν σκεπτικιστές γύρω από αυτό. Και για τον Ντάνιελ, στην τελευταία σας διαφάνεια αναφερθήκατε στην ηγετική συλλογική δράση και στις συλλογικές ε, ε, φιλοδοξίες. Ταυτόχρονα αναφερθήκατε και στα λάθη τα οποία έχουν γίνει και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού ο οποίος δημιουργείται γύρω από το 5G. Τι γίνεται με την Επιτροπή, τι γίνεται με το Κοινοβούλιο, ποιος είναι ο πιθανός ρόλος όλων αυτών των θεσμικών οργάνων. Ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο θα πρέπει να παίξουν και ποιο ρόλο παίζουν σήμερα. Ξέρουμε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να κάνει προτάσεις και το Κοινοβούλιο να οφείσει προς την κατεύθυνση αυτή για τα 5G στο μέλλον. Κούλιτσεκ. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Μία ερώτηση θα έλεγα η ίδια μάλλον και για τους δύο. Βλέποντας τι γίνεται στην Νότια Κορέα, βλέποντας τι γίνεται στην Ιαπωνία, είναι αρκετά επιβλητικές οι εξελίξεις εκεί. Μήπως οφείλεται στο ότι χρησιμοποιούν ένα νέο δίκτυο διαφορετικό από το δικό μας έχουν διαφορετικού τύπου τηλεφωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Μήπως η πρωτοπορία του οφείλεται σε αυτό. Για την δικό μας πυκνότητα του πληθυσμού σχετικά με το 5G χρειάζεται μια υποδομή πολύ πιο πυκνή από αυτή που έχουμε σήμερα ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Και καλά στις πόλεις, εν πάση περιπτώσει, τα μέσα είναι διαθέσιμα, αλλά όταν πηγαίνει κανείς στην Ήπεθρο, στην Νότια Ιταλία, στην, στο νότο της Γαλλίας, στη Γερμανία, στα Καρπάθια, Εκεί υπάρχει μια πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οπότε ίσως όλες αυτές οι εγκαταστάσεις να μην ε, είναι ε, οικονομικά επιθυμητές. Λοιπόν, εδώ έχουν μια κάποια πρωτοπόρο θέση απέναντί μας οι Ιάπωνες και οι Κορέατες, επειδή έχουν επιλέξει ένα διαφορετικό σύστημα και σε ποιο βαθμό απαιτείται υποδομή που να καλύπτει το 100% του εδάφους. Καλώς, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Για τον κύριο Καπόνε, κάποιες ερωτήσεις. Μας έδωσε κάποια στοιχεία ο κύριος Καπόνε για την κατάσταση όπως έχει σήμερα. Υπάρχει ανάγκη από πάρα πολλές υποδομές, υπάρχει ανάγκη από ανάπτυξη τεχνολογιών, υπάρχει ανάγκη για την παροχή νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ολόκληρη σειρά νέων θα έλεγα εφαρμογών είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και την βιομηχανία, τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι προβλέψεις έχετε γύρω από το θέμα αυτό στον τομέα των δημοσίων ε, ε, υπηρεσιών, των δημοσίων τομέων ε, εξυπηρέτησης πολιτών κτλ. Ένα πράγμα είναι οι βιομηχανικές ανάγκες και η ζήτηση, αλλά τι γίνεται για να υπάρξει βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ιδιαίτερα του εργασιακού τους πλαισίου. Προβλέπετε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές εδώ, μήπως υπάρχει δυνατότητα λήψης μέτρων και δημιουργίας τοπικών ας πούμε πλατφορμών, συστημάτων. και να καταλάβω λίγο αυτές οι υπηρεσίες θα είναι υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργούν ε, κερδοσκοπικά ή όχι. Θα αποδίδουν κέρδος ή όχι. Όταν εμείς στο Κοινοβούλιο είχαμε εγκρίνει ε, την απελευθέρωση τμήματος του διαθεσίμου φάσματος, κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο για ορισμένες χώρες, ε, ιδιαίτερα για τον τομέα της αναπετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εντύπωση που είχαμε είναι ότι από πλευρά ορισμένων επιχειρήσεων, ορισμένων χρηστών δεν υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη βιασύνη. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι θέλαμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα. Έτσι προχωρήσαμε στην απελευθέρωση και την πλήρη χρησιμοποίηση του διαθεσίμου φάσματος. Συνεπώς λοιπόν Μιας και υπάρχει κάποιο κόστος ε, με την παροχή τέτοιου τύπου υπηρεσιών, ε, τι ακριβώς γίνεται σχετικά με την πιθανότητα κερδοφορίας της χρήσης αυτών των διαθεσίμων. Και εγώ έχω να θέσω μια ερώτηση, λέει ο κύριος Χένκελ, για τη δοκιμή 5G στο Μιλάνο. Βλέπω ότι με χαρά ότι και συμμετείχε η IBM, η παλιά μου επιχείρηση, στην οποία εργαζόμενα, και επίσης η Q8. Τι ακριβώς γίνεται, τέθηκε το θέμα της προβληματικής της συμμετοχής τέτοιων επιχειρήσεων. Καλώς. Τώρα θα πρέπει να μου δώσουν απαντήσεις ο κύριος Καπόνε πρώτος και ο κύριος Γιώργεφ στη συνέχεια. Ο κύριος Καπόνε θα ξεκινήσω με την ερώτηση τη, σχετική, τη σχετική συγγνώμη με τις επενδύσεις που έθεσε η Ντελ Καστίγιο. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι γενικότερα και ειδικά στην Ευρώπη, αν και γενικά αυτό ισχύει, οι διαχειριστές του δικτύου τα τελευταία χρόνια πιέζονται. Πιέζονται λόγω της μείωσης ε, της, ε, των εσόδων αναχρήστη στο, τον τελευταίο χρόνο. Οι επενδύσεις όμως συνεχίζονται. Έχουν ας πούμε κάνει επενδύσεις στα 4G ε, για διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης και τώρα τους ζητάμε να επενδύσουν για μια νέα υποδομή στο 5G Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις σε ορισμένες χώρες. Μάλιστα το τίμημα του κόστους, μάλλον το κόστος του φάσματος ήταν πάρα πολύ ακριβό. Ε, στην Ιταλία σαν παράδειγμα οι εταιρείε ε, πλήρωσαν 6,5 δις για, την, ε, για το διαθέσιμο φάσμα. Συνεπώς λοιπόν το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό και για τις επιχειρήσεις. Βέβαια σε σχέση με τις αναπτυξιακές τους προοπτικές θα πρέπει να κάνουν ορισμένα προγράμματα και όχι να αναζητήσουν άμεσα την απόσβεση των επενδύσεών τους. Και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα το οποίο ανέφερα προηγουμένως όταν είπα ότι έχουμε να κάνουμε με μια αγορά ιδιαίτερως ανταγωνιστική. Η δημιουργία συνεπώς των προϋποθέσεων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι εταιρείε να μπορούν να προβλέψουν μια κάποια απόσβεση βλέποντας τις πιθανότητες ανάπτυξης των υπηρεσιών έστω και μακροπρόθεσμα. Και χρειάζεται χρόνος εδώ. Όταν αναφερόμαστε σε μια αγορά καταναλωτών Ίσως μερικές φορές ε, είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών. Σχεδόν το 100% του πληθυσμού έχει σε ορισμένες περιφέρειες smartphones και μπορούμε να προβλέψουμε τι έχει να συμβεί με τις νέες υπηρεσίες. Όταν περνάει κανείς το ανεξερεύνητο πεδίο των υπηρεσιών για τις βιομηχανίες, για τις κατασκευές, ε, γενικά ε, τον τουρισμό κτλ τότε θα πρέπει να βρει κάποιες λύσεις. Οι λύσεις λοιπόν αυτές για να βρεθούν απαιτούν επενδύσεις, απαιτούν χρόνο <clears throat> πέρα από την ανάπτυξη απλά των υποδομών. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι περιοχές του κόσμου έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν στις επενδύσεις αυτές. Αυτές οι οποίες θα κινηθούν πρώτες φυσικά και θα εκμεταλλευθούν και θα αναπτύξουν τις λύσεις που απαιτείται. Το θέμα είναι να καταλάβουμε αν η Ευρώπη θέλει να βρει εκ νέου τον βασικό της ρόλο στη πλαίσια της καθοδήγησης ε, του υπόλοιπου κόσμου. Φυσικά είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς και να καθοδηγήσει κανείς τον σχεδιασμό των πολιτικών και του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών που πολλές φορές μεταξύ τους έχουν διαφορές μεταξύ τους. Ακόμα και σήμερα βλέπετε ας πούμε με τις δημοπρασίες φάσματος υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μια κοινή εσωτερική πολιτική. Αναφορικά τώρα με τις δυνατότητες κάλυψης του εδάφους, ιδιαίτερα των περιοχών της υπαίθρου και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν εξακολουθούμε να έχουμε κάποια προβλήματα να κατανοήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτών των επενδύσεων <clears throat> και για τις αστικές περιοχές ακόμα, κατανοείται πόσο πολύ επιφυλακτική μπορεί να είναι ορισμένη για τις περιοχές της υπόθεου. Αλλά υπάρχουν όμως κάποιες υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά και στην Ήπεθρο ε, να επηρεάσουν με δραματικό τρόπο την ε, οικονομία στις περιοχές αυτές, σε όλους τους τομείς, ακόμα και στις περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμιακής. Ε, σκεφτείτε λίγο τον αυτοκινητιστικό τομέα. Δεν μπορείτε να οδηγείτε το αυτοκίνητο μόνο μέσα στις πόλεις και οι υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες να ισχύουν μόνο στην πόλη. Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη ηλεκτρονική και εκτός πόλης. Αλλιώς θα πρέπει να αλλάζει κανείς την οδήγησή του μόνο και μόνο γιατί είναι εκτός κάλυψης. Έρχομαι τώρα στα θέματα των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Τόγια και τις πιθανότητες νέων εφαρμογών. Φυσικά και ο λόγος για τον οποίο γενικά οι πολίτες συγκεντρώνουν την προσοχή τους στα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσει ο βιομηχανικός τομέας από το 5G. <coughs> Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί οι οικονομικές ε, απολαβές θα είναι μεγαλύτερες. Αλλά φυσικά και ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ένας από τους τομείς στους οποίους μπορεί να αναμένει κανείς πάρα πολλά πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά νέου τύπου από το 5G. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να κατανοήσετε καλύτερα που βρισκόμαστε. Ένας από τους τομείς στους οποίους πιστεύω ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να ωφεληθεί ιδιαίτερα από την προχωρημένη αυτή συνδεσιμότητα είναι ο τομέας της υγείας. Σαν παράδειγμα, συνδεδεμένα νοσοκομιακά οχήματα. Μπορούν να αλλάξουν εντελώς την μορφή της κατεπίγουσας βοήθειας. Εδώ ο χρόνος είναι το βασικό, το καθοριστικό χαρακτηριστικό. Και αν μπορεί κανείς σαν παράδειγμα ε, να ξεκινήσει την φροντίδα του ασθενού στο εσωτερικό του νοσοκομιακού οχήματος, έχοντας τον ασθενή συνδεδεμένο με τα κεντρικά στελέχη ε, του νοσοκομείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης του τραυματία, σαν παράδειγμα, ή του ασθενούς. Αλλά επίσης μπορεί να υπάρξει και μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσιών της Ευρώπης, γιατί κάποιοι μπορούν να μένουν στο σπίτι τους και να παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, να είναι συνδεδεμένοι και όχι να είναι στο νοσοκομείο. <clears throat> Συνεπώς λοιπόν ακόμα και η ποιότητα ζωής την οποία θα έχουν τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα θα βελτιωθεί με δραματικό τρόπο. Με πολύ σημαντικό τρόπο διότι θα παραμένουν διασυνδεδεμένοι με τις κεντρικές μονάδες υγείας. Ο τομέας ο δικός μου, η εκπαίδευση και εδώ μπορεί να υπάρξει όφελος ιδιαίτερο από το 5G. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η νέα γενιά, οι ε, φοιτητές μας ε, λειτουργούν διαδραστικά <clears throat> με διαφορετικό τρόπο με τον οποίο το κάναμε εμείς, η δική μου γενιά. Δεν είναι ότι είναι διαφορετικοί οι ίδιοι, αλλά ο τρόπος δράσης τους είναι διαφορετικός. Συνεπώς λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι νέες γενιές είναι και αυτός διαφορετικός. Πρέπει να προσαρμιστούμε στο νέο τρόπο εκπαίδευση λοιπόν και να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση σε αυτό τον νέο τρόπο πρόκλησης κοινωνικής αλληλοεπίδρασης και κοινωνικής διαδραστικότητας. Νομίζω ότι εδώ η προχωρημένη συνδεσιμότητα μπορεί να βοηθήσει τις κοινότητες οι οποίες ακόμα και αν δεν έχουν φυσική επαφή να συνδέονται, να συνδέονται οι φοιτητέ μεταξύ τους, να συνδέονται οι φοιτητέ με τους καθηγητές τους κτλ. Και τέλος, οι λεγόμενες ευφυείς πόλεις. Μιλάμε γι' αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες ε, τις οποίες έχουμε ήδη αναπτύξει στις πόλεις είναι η έλλειψη ε, διαθέσιμης και ευθυνής συνδεσιμότητας. Ευτυχώς πολλές από τις υπηρεσίες αυτές που μπορεί να έχει καλύπτονται από το 5G και μία από τις προκλήσεις του 5G είναι η προσαρμοτικότητά του. Θα ήθελα να πω ότι όταν αναφέρεται κανείς τις ευφυείς πόλεις ή τις υπηρεσίες διαδικτύου των πραγμάτων, στην ουσία αναφέρεται κανείς σε συνδεσιμότητα χαμηλής ταχύτητας, low rate connectivity. Δεν είναι όμως ο μόνος τρόπος που πρέπει να δει κανεί αυτές τις υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες και η διάδρασή μας με τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες γίνεται μέσω μιας οθόνης. Δεν πρέπει όμως να γίνεται μόνο με απεικονιστικό τρόπο. Οι υπηρεσίες στα πλαίσια του εφιούς περιβάλλοντος δεν μπορούν να γίνονται μόνο μέσω στενού φάσματος, δηλαδή στην ουσία να υπάρχει ένα link, ένα σύνδεσμος ανάμεσα στα διαφορετικά σημεία σώρευσης ή φύλαξης δεδομένων. Μπορεί να υπάρξει και σύνδεση ευρέως φάσματος που να επιτρέπει τη μη χρήση, σαν παράδειγμα, της οθόνη ενός κινητού ή ενός άλλου, μιας άλλης πλατφόρμας. Αυτό θα δημιουργήσει το λεγόμενο FES περιβάλλον. Um, ο κ. Γκιόργεφ. Όταν μου ζητήθηκε να συντομεύσω την παρουσίασή μου στα 10 λεπτά, χρειάστηκε να αφήσω εκτός κάποια πράγματα και χαίρομαι που μου ετέθη το ερώτημα. Αν δούμε την RSPG και να δούμε το έργο που έγινε κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρία και της προηγούμενης, ε, ε βλέπουμε ότι αρχίζουμε και βλέπουμε τους καρπούς της ε, στενή συνεργασία. Εμπειρογνώμονε ειδικοί από διάφορε χώρες συναντώνται και εξηγούν γιατί κάνουν αυτό που κάνουν όπω το κάνουν και μοιράζονται τις καλύτερε, τις βέλτιστε πρακτικές. Και αυτό νομίζω θα βοηθήσει στην επιτυχία της, ε, των δικτύων πέμπτης Γενιά στην Ευρώπη. Το γεγονό ότι τα δύο όργανα θα συνεργαστούν ε, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Γιατί όλες οι προκλήσεις οποίες ανέφερα, την ανάπτυξη του δικτύου, το φάσμα κλπ, όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών πλέον. Οπότε πρέπει συνεχώς να οθούνται και να ενθαρρύνονται να προχωρήσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους εξαιτία τη φύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου δεν είναι μία μοναδική χώρα, επειδή περιλαμβάνει 28 κράτη-μέλη, χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία και το συντονισμό για να ανταγωνιστούμε με μεμονωμένες χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η, η, η Κίνα. Τώρα για την Κορέα. Κύριε Κολτσεκ, έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Η Νότια Κορέα είναι ένα από τα πιο καλά παραδείγματα ε, ταχείας ανάπτυξης των δικτύων πέμπτης γενιάς και έχουν και το, πλεόνας, το πλεονέκτημα ότι έχουν μικρό πληθυσμό, είναι μικρή χώρα οπότε μπορούν να προχωρήσουν και πολύ πιο γρήγορα έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Μέχρι το 2025 θέλουν να καλύψουν το 60% με συνδέσεις πέμπτης γενιάς. Οπότε είναι πάρα πολύ ρεαλιστέ σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Πέρσι ε, ε, δημοπράτησαν συχνότητες μιλιμετρικές καθώς επίσης και τη C-band ε, και έδωσαν ο, 800 ε, MHz σε κάθε ε, στους παρόχους μιλιμετρικών συνδέσεων. Κάνουν λοιπόν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τα ενία. Και αυτό είναι που, που διακρίνει αυτή η χώρα. Τώρα, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει δύο βήματα πιο πίσω. Έχουμε 28 κράτη-μέλη που πρέπει να συνεργαστούν καταρχήν. Και έχουμε και προκλήσεις που δεν έχει η Νότιος Κορέα. Για παράδειγμα, το ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις πόλεις και τις αγροτικέ περιοχές. Οπότε, έχουμε αυτό το μειονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα αυτό το μειονέκτημα καθιστά αυτή την τεχνολογία πιο ελκυστική από ό,τι στην Νότια Κορέα. Οπότε θα πρέπει η Ευρώπη να επιδείξει μια βούληση συνεργασίας και συλλογικής ηγεσία. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ξεκι... Προχωράμε στην δεύτερη συνεδρία. Θα συζητήσουμε το ρόλο των ε, ε, ε, των δορυφόρων στην, στα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανιέλη, διευθυντή των θεσμικών ε, θεμάτων της ε, UTELSAT και θα μας ε, παρουσιάσει ε, τις δορυφορικές ε, τεχνολογίες και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της πέμπτης γενιάς. Ο κύριος Ανιέλη δεν έχει σχέση με την οικογένεια Ανιέλη, πρέπει να σα το πω αυτό γιατί ξέρω ότι θα έχετε όλη την περιέργεια. Δέκα λεπτά κύριε Ανιέλη. Πράγματι, δεν είμαι συγγενής του πρώην ιδιοκτήτη της Fiat. Θα σας μιλήσω όχι μόνο για το ρόλο των δορυφόρων στην πέμπτη γενιά, αλλά συνολικότερα το ρόλο των δορυφόρων στην συνδεσιμότητα του ψηφιακού μέλλοντος. Θα μιλήσω για την ε, αλυσίδα, αλυσίδα αξίας και τα, τις μελλοντικές τάσεις σε σχέση με τους δορυφόρους. Δεύτερον, ε, ο ρόλος των ε, δορυφόρων για την γεφύρωση του, της δια, διαφοράς και μετά η ενσωμάτωση του 5G με το ίντερνετ, το ίντερνετ των πραγμάτων. Τέλος θα βγάλω κάποια συμπεράσματα. Καταρχήν να σας πω πού που, που, που, έρχομαι, ποιο είναι το δικό μου πανόραμα. Εδώ εκπροσωπώ τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Έχουμε τους ε, κατασκευαστές, ε, ε, τους, τις εταιρείες που στέλνουν δορυφόρους στο διάστημα, τους εκτοξευτές δηλαδή. Το μέσον έχουμε τους παρόχους και εδώ θέλω να σας πω ότι στην Ευρώπη έχουμε ηγετικέ εταιρείε. Είμαστε ηγέτες στον τομέα των ε, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και των αντίστοιχων εμπορικών παρόχων. Είναι πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι εταιρείε. Ε, μεταξύ αυτών η Eutelsat. Να σας δίνω και δυο και μερικά νούμερα για την Eutelsat. Το σημαντικό είναι ότι οι πάροχοι ε, δορυφορικών υπηρεσιών ε, είναι στην πραγματικότητα πάροχη υποδομών. Τίποτα άλλο, σύμφωνα με τον καινούριο κώδικα. Αν έπρεπε να μόνο, να, να θυμηθείτε μόνο μία φράση, είναι ότι ο τομέας των δορυφορικών επικοινωνιών εξελίσσεται. Και τεχνολογικά και επιχειρηματικά. Αυτή η εξέλιξη αφορά και τον συμβατικό κλάδο των σταθερών ε, συνδέσεων ε, αλλά και πιο προς ε, σύγχρονους τομείς όπως η κινητή τηλεφωνία και οι κινητές συνδέσεις. Οι δορυφορικές επικοινωνίες μπορούν να φέρουν άνευ φόρων και άνευ περιορισμών συνδεσιμότητα παντού μεταξύ αυτών και στο, στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές εκτός πόλεων. Οπότε μέσω, αυτών, μέσω αυτής της μπορούμε να διαθέσουμε πάρα πολλές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σύνδεση με πλοία, σύνδεση με αεροπλάνα, συνδεσιμότητα σε περιπτώσεις ε, θεομηνιών, όλα αυτά ε, μπορούν να λάβουν χώρα μόνο μέσω δορυφορικών συνδέσεων και επικοινωνιών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δορυφόρων. Πρώτον, ευρία κάλυψη και παρουσία παντού. Επίσης όμως και ε, αποτελεσματική σε ό,τι αφορά το κόστος, ε, μετάδοση υπηρεσιών ε, διανομής περιεχομένου σε υψηλές ταχύτητες. Η, η χρήση των δορυφόρων μπορεί να συμπληρώσει άλλα δίκτυα ε, για, και για την ε, παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης, ε, κινητών δικτύων, κινητής τηλεφωνίας, αλλά αργότερα και ίντερνετ των πραγμάτων κλπ. Το ψηφιακό χάσμα. Ψηφιακό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλου τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020, το ψηφιακό χάσμα εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Δέστε για παράδειγμα την κάλυψη 30 Mbit per second, που θα υποτίθεται θα πρέπει μέχρι το 2020 να είναι διαθέσιμο σε όλους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80%. Καλύπτουμε μόνο το 80% του πληθυσμού. Πάνω 50 εκατομμύρια δηλαδή άτομα είναι εκτός αυτής της κάλυψης. Πιο σημαντικό όμως. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται στις αγροτικές περιοχές. Μόνο το 50% αυτών ε, έχουν ε, ευρεία ευρυζωνική σύνδεση και μόνο το και 8% ε, δεν καλύπτεται καν. από διαδικτυακή σύνδεση. Και μάλιστα μπορεί ποτέ να μην καλυφθούν, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δύσκολη η πρόσβασή τους. Τώρα, έχουμε και τον καινούριο κώδικα, τους στόχους της κοινωνίας του Gigabit. Όμως, η συνδεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται πολύ των στόχων του 2020. Οπότε, αν χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αριστοτέλη, η πρόοδος δεν αξίζει τίποτα εκτός και αν αφορά όλους. Ή για να το πω με τα λόγια του Βολτέρου, είναι το καλύτερο εχθρός του, κακού, του καλού. Προηγουμένως αναφέραμε τον, το, τη λέξη φιλοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, χρειάζεται να συνδυάσουμε τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ηγηθεί της ψηφιακής οικονομίας με την επίγουσα ανάγκη να συνδεθούν όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερως σε αγροτικές περιοχές, στο ίντερνετ. Μην ξεχνάμε ότι οι αγροτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 20% πάνω από το 20% του πληθυσμού. Εδώ μπορούν να βοηθήσουν οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες διότι μπορούν να συμπληρώσουν τις, ε, τη συνδεσιμότητα σε περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται ή υποεξυπηρετούνται και με, ένα, με μια μικρή επένδυση ανανοικοκυριών ανεξαρτήτως της θέσης του. Και οι υπάροχοι τέτοιων υπηρεσιών κάνουν επενδύσεις και θα, φέρουν, θα αυξήσουν την ε, παροχή υπηρεσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Το καλό είναι ότι αυτές οι επενδύσεις δεν θα καλύπτουν μόνο πληθυσμό, αλλά και επικράτεια και κόστος και τις θάλασσες και τις ε, ε, πιο σημαντικές ε, διαδρομές αεροπλάνων. Και όπως σας είπα, οι δορυφόροι εξελίσσονται το ίδιο και οι ικανότητές τους, οι επιδόσεις τους. Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και το έδαφος αλλά και στον ουρανό. Αυτό μας φέρνει στην πέμπτη γενιά. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ξανά το τρίγωνο. Μας το εξήγησε ο κύριος Καπώνη αρχικά. Αλλά το σημαντικό είναι οι υπηρεσίες πέμπτης γενιάς να καταστούν διαθέσιμες παντού. Και αυτό αποτελεί πραγματικά πρόκληση. Προκειμένου δηλαδή να καλυφθεί καλυφθεί όλη η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πέμπτη γενιά. Και είναι σημαντικό να καλύψουμε όχι μόνο πληθυσμό, αλλά και γη και έκταση. Επικράτεια. Οπότε η, στο μέλλον η επιτυχία της πέμπτης γενιάς θα εξαρτηθεί από το πώς θα συνεργαστούν σωστά ε, στις προσπάθειές τους διάφοροι πάροχοι. Καμία τεχνολογία από μόνη της δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ε, δηλαδή υψηλή ταχύτητα σε πολύ, με πολύ χαμηλή ε, καθυστέρηση και για χιλιάδες τέρμιναλ, ε, τελικούς χρήστες δηλαδή. Όμως, το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογίες και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αρκετά ευφυές έτσι ώστε κάθε φορά να χρησιμοποιεί τη σωστή τεχνολογία για τον κατάλληλο χρήστη και τις κατάλληλες εφαρμογές. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ποιες είναι οι, οι, οι, οι χρήστες στρατηγικής χρήσης. Ε, Γιατί, γιατί οι τεχνολογίες αυτές μπορούν, η τεχνολογία αυτή μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το χρήστη, με τρόπο διαφανή. Οπότε, οι φιλοδοξίες μας για την πέμπτη γενιά έχουν ανάγκη και τους δορυφόρους. Χρειάζεται τα δίκτυα να πυκνώσουν, σίγουρα. Αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στα δίκτυα οπτικών ινών. Χρειάζεται να επιλέξουμε ένα μείγμα τεχνολογιών. Και οι δορυφόροι, από αυτή την έννοια, προφανώς δεν είναι κατάλληλοι για όλε τι υπηρεσίες. Είναι όμως εξαιρετική επιλογή για ένα αριθμό υπηρεσιών. Εκεί όπου χρειάζεται, για παράδειγμα, ταχύτατη ε, σύνδεση. Εκεί που χρειάζεται να συνδέσουμε ε, κόμβους σε, στην ύπεθρο. Ή κινητούς κόμβους, για παράδειγμα αεροπλάνα ή πλοία εκεί όπου χρειάζεται, εκεί που είναι κατάλληλο κάθε φορά. Γιατί το δίκτυο θα είναι αρκετά ευφυές έτσι ώστε να επιλέγει την κατάλληλη οδό, την κατάλληλη τεχνολογία για να φτάσει στο χρήστη. Το ίντερνετ των πραγμάτων. Εντάχει. Και εδώ λέξη κλειδί είναι η ολοκλήρωση με τα χερσαία δίκτυα και η ε, παρουσία παντού. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής της τεχνολογίας, δορυφορικής τεχνολογίας στο ίντερνετ των πραγμάτων. Κοιτάξτε, προσέξτε τι, τι πρέπει να προσέξουμε εδώ. Οι δορυφόροι θα εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους, τα ίδια αντικείμενα ε, και θα στέλνουν τα ίδια μηνύματα, θα χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες με τα χερσαία δίκτυα. Οπότε η ολοκλήρωση όχι μόνο είναι δυνατή, αλλά είναι και απαραίτητη. Τώρα, συμπεράσματα. Οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες φέρνουν διευρυμένη κάλυψη και παρουσία παντού, καθώς επίσης και παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας αποτελεσματικά και με σχετικά χαμηλό κόστος. Διευρυμένη κάλυψη σημαίνει επίσης ότι πολεμάμε με αυτόν τον τρόπο και το ψηφιακό χάσμα που αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη. Επίσης, σημαίνει ότι μπορούν οι δορυφόροι να χρησιμοποιηθούν για ταχεία ανάπτυξη σύνδεση σε συνεργασία και συμπληρωματικά των χερσαίων υπηρεσιών. Και βέβαια οι δορυφόροι επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή του ίντερνετ των πραγμάτων ε, ε, σε συνεργασία πάλι με τις χερσαίες τεχνολογίες. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια όρεξη σε αυτούς που ζουν στην... Ε, να ανοίξουμε την όρεξη σε αυτούς που ζουν στην Ήπεθρο. Δεν μπορούμε να τους πούμε ότι θα περιμένουν 10 χρόνια να αναπτυχθεί το χερσαίο δίκτυο λοιπά και μετά να αρχίσουν οι επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βιαστούμε και οι δορυφόροι μπορούν να, χρησιμοποιη... να χρησιμεύσουν εκεί. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε δηλαδή την εισαγωγή του ε, ε, ευρυζωνικού ίντερνετ στην Ήπεθρο. Τέλος, δεν υπάρχει κανός είδους δικαιολογία για να μην εξασφαλίσουμε ψηφιακή συνδεσιμότητα σε όλους. Συστάσεις. Προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την συμπερίληψη της δορυφορικής ε, επικοινωνίας στις ε, πολιτικές που επεξεργαζόμαστε Πρώτον, για να καταπολεμήσουμε το ψηφιακό χάσμα και δεύτερον, για να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση του ε, των ευρυζωνικών υπηρεσιών πέμπτης γενιάς και των υπηρεσιών πέμπτης γενιάς. Αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν παράλληλα. Οι δορυφορικές επικοινωνίες ε, δίδουν μια επαρκή υποδομή για να στηρίξουν ευρωπαϊκές πολιτικές και κρίσιμη υποδομή σε στιγμές κρίσης. Τέλος, ό,τι αφορά την βιομηχανική πολιτική, μην ξεχνάμε ότι η SATCOM είναι ένα τμήμα μιας συνολική αλυσίδας αξίας. Ε, επενδύει ο τομέας στην ευρωπαϊκή ε, τεχνολογία, κάτι που είναι σημαντικό ε, για την ανταγωνιστικότητα του συνολικού ε, τομέα της αεροβιομηχανίας στην Ευρώπη, Airbus, Thalys κλπ. Και η Utelsat επίσης είναι ε, και πολύ καλό μας πελάτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανιέλη. Παρακολουθώντας την ε, ομιλία σας μου ήρθε μια ιδέα. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα μητροπολιτικά κέντρα γίνονται όλο και μεγαλύτερα και δύσκολα να τα διαχειριστεί κανείς και μεγάλα τμήματα εγκαταλείπονται Ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε ανάποδα, δηλαδή να βάλουμε το 5G στην Ήπεθρο πρώτα. Τώρα, ο κύριος Μάρτιν Μπόργεσον, παρακαλώ να λάβει τον λόγο, θα ομιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη, τις εφαρμογές της και τα 5G. Ορίστε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Είναι σημαντική η τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ ενώπιον σα σήμερα. Η παρουσίασή μου θα είναι λίγο διαφορετική. Θα αρχίσω με μια ερώτηση και μετά θα μιλήσω λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη και ιδίω βέβαια σε συνδυασμό με το 5G. Και θα έρθουμε μετά στι ερωτήσει. Ελπίζω ότι θα εξυπηρετήσω έτσι τους σκοπούς σας. Λέγομαι Μπόργεσον και είμαι εταίρο στην 2021.ai, αλφαγιώτα, στην Κοπενχάγη και έχω ε, ένδον γνώση την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και πρώτα σε ό,τι αφορά την διασυνδεσιμότητα και το 5G υπάρχει μια ερώτηση που έρχεται στα χείλη μου και ας πούμε ότι εγώ επιθυμώ να δωρήσω τα προσωπικά μου δεδομένα και τα οικογενειακά μου δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μου, τη Σουηδία, στην περιφέρειά μου και στον τοπικό δήμο, στην κοινότητα όπου ζω και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό. Για να τα δωρήσω αυτά χρειάζεται διασυνδεσιμότητα. Δεν τα λέω αυτά διότι είναι μια ανοητή ιδέα, αλλά διότι θα δημιουργούσε αυτό τεράστιες ε, δυνατότητες για όλους αυτούς τους φορείς να συμβάλλουν στην βελτίωση της κοινωνίας. Μια κοινωνία πιο ευχάριστη για να ζει κανεί και που να μα επιτρέπει και να δορίζουμε τα δεδομένα αυτά για το καλό τη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αρχίσουμε να τα σκεπτόμαστε αυτά, ακόμα και αν έχουμε αρχίσει να σκεπτόμαστε και άλλα πράγματα, δηλαδή πώ θα αντιμετωπίσουμε το άτομο μέσα στα πλαίσια τη διασυνδεσιμότητα. Και αν προχωρήσουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, στην παγκόσμια οπτική, υπάρχει εδώ μια εικόνα που ίσως είναι κάπω αρνητική Πάντω δείχνει ότι υπάρχει κάποιο δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να εκτιμηθεί. Πρώτα, δεν είμαστε μεταξύ των χωρών που ηγούνται τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχουμε ούτε την ικανότητα, ούτε μια ξεκαθαρή στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε έχουμε και τους ε, απόλυτα ικανούς φορείς στα πανεπιστήμια και δεν έχουμε και ευρύτερη συλλογή δεδομένων. Αν δείτε τις διάφορες χώρες θα δείτε ότι σαφώς σήμερα οι Κινέζοι προηγούνται, οι ΜΟΝ, έχουν δύο βασικά θετικά στοιχεία, προς το με παρεξηγήστε, αφενός έχουν 1,4 δισεκατομμύρια Κινέζους πολίτες, σε ό,τι αφορά δε τις εταιρείε τους, και βεβαίως εκεί κινούνται Facebook και Instagram και εκεί συλλέγουν τα δεδομένα. Υπάρχει στρατηγική τέχνη τη νοημοσύνη κινέζικη, υπάρχει και ρωσική. Πάλι μην με παρεξηγήσετε, αλλά δεν νομίζω ότι εμεί έχουμε επί του παρόντο στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και να μα δείχνει που θέλουμε να κατευθυνθούμε σε θέμα τεχνητή νοημοσύνης. Ούτε καν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν στρατηγική τεχνητή νοημοσύνη. να φτιάξω ένα τείχο, το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ αποτελεσματικό. Και α επανέλθουμε στα δεδομένα και επανέρχομαι σε αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά. Γιατί είναι ένα τομέα όπου πρέπει να φτιάξουμε και να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις μοιραστούμε για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες μιλήσαμε. Για παράδειγμα στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, στις ευφυείς πόλεις και στις ευφυείς υποδομές. Όλα αυτά πρέπει να βασιστούν σε δεδομένα. Άρα πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί το θέμα αυτό της συλλογή δεδομένων. Αυτό βεβαίως δεν είναι και δωρεάν. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πρώτα να θεσπιστούν. Έχω το, ε, το ακρόνιμο MELTS που σημαίνει mindset, δηλαδή νοοτροπία, διανοητική διάθεση. Για παράδειγμα για την η φροντίδα της υγείας, προληπτική. Εκεί πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και ε, να συλλεχθούν πάρα πολλά δεδομένα. Ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε μετά στον πειραματισμό, experimentation. Να αναλάβουμε καλά υπολογισμένους κινδύνους, ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Χρειαζόμαστε ικανή ηγεσία, leadership, πάλι μετρημένη με τους κινδύνους και εκεί χρειάζεται μια πολύ ε, λεπτή ισορροπία. Ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Αλλιώ θα χάσουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε μια πραγματική ψηφιακή ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλο, χρειαζόμαστε δεδομένα, data, το D στο MELTS και χρειαζόμαστε και δεξιότητε, το S skills του MELTS και να εκπαιδεύσουμε επαρκεί αριθμού επιστημόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ικανοποιηθούν οι ανάγκε του μέλλοντο. Και αυτοί θα ωφελήσουν όλες τις βιομηχανίες, ιδίω όμως θα ε, εξυπηρετήσουν το κοινό, το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει τις ανάγκες και εκεί θα πρέπει να ισχύσει αυτό το μήνυμα που περιλαμβάνει στο ακρόνιμο MELTS. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική. Η στρατηγική δεν χρειάζεται να είναι και ιδιαίτερα περίπλοκη. Αν βγάλουμε την πλευρά του business, που γι' αυτό μιλώ συνήθως στους επιχειρηματίες. Χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή κοινωνία. Ας προχωρήσουμε σε αυτό. Και νομίζω τότε θα μπορέσουμε ε, να δημιουργήσουμε στρατηγικά asset, τα οποία δεν έχουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε ικανότητες χρειαζόμαστε και ελέγχους. Έχουμε αρχίσει από τους ελέγχους. Διοντολογική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί δηλαδή πάμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο ελέγχων. Αλλά δεν έχουμε βάλει στόχους και η διασυνδεσιμότητα θα αποτελέσει θεμέλιο για τη στρατηγική αυτή, διότι αν δεν υπάρχει διασυνδεσιμότητα δεν θα μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα. Και αν δεν μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα, δεν μπορείτε και να τα χρησιμοποιήσετε και να φτιάξετε μια καλύτερη κοινωνία στη βάση τους. Να λοιπόν η διασυνδεσιμότητα και το 5G, το οποίο 5G θα μεταμορφώσει σιγά σιγά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες όχι μόνο ιστορική πληροφορία, δηλαδή αυτή που αναφέρει στο παρελθόν, αλλά και τρέχουσα. Και μιλούμε για αισθητήρε. Εγώ έχω ένα αισθητήρα στον βραχιονά μου και τελικά νομίζω όλοι θα έχουμε αισθητήρε μέσα μα, στο σώμα μα, που θα βελτιώνουν την ανθρωπιά μα και θα μα λένε πότε πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, για παράδειγμα. Και θα μα το λένε ακριβώ τη συγκεκριμένη στιγμή που πρέπει. Εγώ νομίζω ότι θα είναι καλό, διότι θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τότε την ε, ε, ζήτηση και όχι να ξεκινούμε από την προσφορά. Τέλος, η κινητικότητα στην υγεία. Δεν έχω τώρα τα business case μαζί μου, μπορούμε να υπολογιστούν τα πράγματα αυτά. Υπάρχει όμως μεγάλη συμφωνία και βούληση να εξεταστεί αυτό. Ήδη οι ιδιωτικοί φορείς το κάνουν αυτό. Πιστεύω όμω ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκύψει, διότι μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα αυτά καλύτερα, ευφιέστερα, μέσω τη διασυνδεσιμότητας, αλλά και με συλλογή δεδομένων. Επανέρχομαι στην ερώτησή μου λοιπόν. Μπορείτε να με βοηθήσετε, μπορείτε να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο με τη διασυνδεσιμότητα 5G, αλλά και με τη συλλογή των δεδομένων. Εγώ θα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο αν μπορείτε να με βοηθήσετε να δωρήσω, όπω είπα, τα δεδομένα μου σε διάφορου φορεί που θα τα χρησιμοποιούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και Μπόργεσον σε ό,τι αφορά την δωρεά δεδομένων. Εμένα πάντως με πείσατε. Ίσως όμως να είμαι και ο μόνος μεταξύ των 751 ευρωβουλευτών που επίστη. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου ενδιαφέρονται τόσο πολύ για προσωπική σφαίρα και διάφορα αυτά. Ερωτήσεις τώρα κύριε και κύριοι. ask uh, a question on this uh, privacy. από το θέμα της ιδιωτικότητας, τι θα συμβεί αν όλοι δώσουν όλα τα προσωπικά τους δεδομένα έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να έχει και αυτός πρόσβαση σε ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας την τεχνητή μου ημοσύνη για να βρει καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες της κοινωνίας. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αποδεκτό. Κοιτάξτε, είναι μια ιδέα, ως εκ τούτου μπορεί να μετασχηματίσει ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία υγείας, ας πούμε, για την έβρεση και χρήση των σωστών φαρμακευτικών ουσιών. Νομίζω ότι η δημοκρατία όμως πρέπει να είναι το θεμέλιο στη συλλογή και επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Εγώ έχω κάποια καρδιολογικά προβλήματα και ο καρδιολόγος είπε ότι θα μπορούσε να μου φυτέψει κάτι έτσι ώστε αν υπάρξει ένα πρόβλημα να ενημερωθεί μέσα από το iPhone μου αυτόματα και να μου τηλεφωνήσει και να μου πει θα κάνω αυτό ή το άλλο που ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί ασθενείς με τέτοιου είδους ε, αισθητήρε εμφυτευμένους, συνεπώς δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι και το τρομερά δραματικό και καινοτόμο. Όχι, σύμφωνο. Απλά θεωρώ ότι, ότι ίσως πρέπει να περιμένουμε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την αποδοχή αυτών των διαδικασιών. Όταν κάποιος πρέπει να κάνει μια τέτοια εμφύτευση απαιτείται μια κάποια εμπιστοσύνη. Από την άλλη αυτό θα ήταν καλύτερο εφόσον η ζωή μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα ζητήσω από τον κύριο Στούκμαν, από την Γενική Διεύθυνση Connect, να κάνει κάποιες παρατηρήσεις και κάποια συμπεράσματα από τις συζητήσεις μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις και για μας Εμείς εφαρμόζουμε το πρόγραμμα δράσης 5G σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα εκλεκτά μέλη, τα οποία μας βοήθησαν να καθορίσουμε τους κανόνες τους εφαρμοστέους στα πλαίσια της 5G Το πρόγραμμα δράσης 5G ε, είναι κάτι το οποίο στηρίχθηκε πάρα πολύ από το σώμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ να προχωρήσουμε στην ε, πολι... τη χάραξη της πολιτικής. Και το παρατηρητήριο για την ε, για τα θέματα αυτά επίσης βοηθήθηκε στην εκκίνησή του και στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος πενταετούς δράσης. Βλέπουμε ότι πράγματι σε επίπεδο δοκιμών η Ευρώπη βρίσκεται σε μια ηγετική θέση. Έχουμε μεγάλης κλίμακας δοκιμές στην Ευρώπη και στα πλαίσια της χρηματοδότησης του προγράμματος που ε, εμείς αναπτύσσουμε σε, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και σε πολλά από τα προγράμματα αυτά συμμετέχουν φυσικά και δορυφόροι. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα, υπάρχει η πολυδιάσπαση της αγοράς, όπως είπατε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν είμαστε πρώτοι οι οποίοι θα αναπτύξουμε τις νέες αυτές αγορές και σε σχέση με τη χρήση του φάσματος Νομίζω ότι το 10% επιπλέον φάσματος και στα τρία επίπεδα στις τρεις κατηγορίες θα πρέπει να αποδοθεί μέχρι το 2020. Συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Αλλά έχουμε νομίζω τα απαιτούμενα μέσα τα οποία θα μας επιτρέψουν να προχωρήσει η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενθαρρύνουμε για την επίτευξη των στόχων όπως είπαν και οι πανελίστες. Καταρχάς η δημιουργία των λεγόμενων οικοσυστημάτων είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε και το κάνουμε. Το 5G δεν είναι μόνο κατανάλωση, είναι κάθετες επιχειρηματικές προσπάθειες, ε, κάποιοι από σας ε, τα ε, έκαναν την περιγραφή. Σαν παράδειγμα, συνδεδεμένη ή διασυνδεδεμένη κινητικότητα, η κυρία Γκάμπριελ σαν παράδειγμα συνεργάθηκε με τους συμμετέχοντες στην αγορά για την ανάπτυξη των συστημάτων για την αυτοκίνηση. Έχουμε και τις προτάσεις τις οποίες υποστηρίζει το Κοινοβούλιο. Θέλουμε λοιπόν εμείς στα πλαίσια του Connected Europe να βοηθήσουμε και τα προγράμματα ανάπτυξης έτσι ώστε να επιταχύνει η Ευρώπη. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, και σε σχέση με τις λεγόμενες κάθετες παροχές υπηρεσίας την επόμενη δεκαετία. Υποστηριζόμεθα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα για το ίντερνετ των πραγμάτων και το 5G υπάρχουν ε, μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα. Το ίντερνετ των πραγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στα δίκτυα αυτά. Έχουμε ήδη μια στρατηγική από πέρυσι όπου είδαμε ποιες είναι, αναζητήσαμε τις ευκαιρίες τις οποίες μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, όπως επίσης και τους κανόνες σε επίπεδο δεοντολογίας για να γίνουν οι υπηρεσίες αυτές, ε, θα έλεγα, αξιόπιστες. Σχετικά με τις δημοσιονομικές προτάσεις, εμείς έχουμε πλέον την δυνατότητα να συνεργαστούμε σε εταιρικέ σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα και με το Internet of Things. Τώρα, ε, στην ερώτηση Μάρτιν. One of our priorities under Horizon Europe, that's also one program that is Για την δωρεά των δεδομένων, αυτό είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε ένα ανθρωποκεντρικό διαδίκτυο, αυτό έχει σημασία. Και εδώ νομίζουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι χώροι προσωπικών δεδομένων, δεν είναι ακόμα έτοιμοι βέβαια. Θα ξεκινήσουμε στα επόμενα προγράμματα γύρω από αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήνουμε τον χρήστη να αποφασίζει για το αν μπορεί να εντάξει τα δεδομένα του ε, σε ένα σύνολο δεδομένων, σε μια δέσμη δεδομένων και ποιος θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης. Μπορεί να επιτρέπει την χρήση των δεδομένων του ελέγχοντάς τα όμως. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς σας ζητούμε να στηρίξετε τα ψηφιακά προγράμματα. Μόλις συνειδητοποίησα ότι ο κύριος Καπένε, Καπόνε συγγνώμη, δεν μου απάντησε ακόμα στην ερώτηση που έκανα για την συμμετοχή της Huawei στα πειράματα στο Μιλάνο. Ε, ε, well, the, the, ε, the trial in Milano is based on full coverage of the metropolitan. Λοιπόν, αυτό καλύπτει το σύνολο της Μητροπολιτικής Περιοχής ε, του Μιλάνου, 300 site και τα μισά από αυτά τα παρέχει η Huawei. Έχει μοιραστεί η πόλη λοιπόν σε δύο μέρη και το ένα καλύπτεται από τα μέσα τα τεχνικά της Huawei. Εμείς ε, δεν είχαμε κάνει τέτοιες συζητήσεις ε, ε, στα πλαίσια του καθορισμού της δοκιμής ε, συνεργασίας με την Huawei. Θα πρέπει να πω όμως ότι από αυτά τα οποία βλέπω στην παρούσα φάση, το επίπεδο επένδυσης στην έρευνα από την Huawei είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτή είναι όμως η προσωπική μου άποψη, ενός ακαδημαϊκού, ενός πανεπιστημιακού ο οποίος ενδιαφέρεται να υπάρχουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και στην έρευνα. Στην παρούσα φάση λοιπόν αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι το επίπεδο το επενδυτικό το οποίο προέρχεται από την Huawei και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον τηλεπικοινιακό τομέα, αλλά η Κίνα γενικά επενδύει και αυτό δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα έρευνα στα οποία στα οποία επενδύει η Ευρώπη, τουλάχιστον σε εταιρικό επίπεδο. Γιατί σε επίπεδο δημόσιων επενδύσεων ξέρουμε, ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρισκόμαστε. Δεν ε, βλέπω λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε ε, και νομίζω ότι οι παίκτες οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν στην ανάπτυξη συστημάτων 5G στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ λίγοι. Προφανώς θα πρέπει να εξισορροπήσουμε ακόμα περισσότερο τις ανησυχίες που έχουμε και για επενδύσεις με τις ανησυχίες με τα θέματα της ασφάλειας. Καλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές λοιπόν για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους και τις ε, εξαιρετικές απαντήσεις και ερωτήσεις. διαχειριστήκαμε την συζήτηση με εξαιρετικό τρόπο και θα συναντηθούμε εκ νέου στις 4.30. Ρικομβίνια.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 Okay, ladies and gentlemen, now <clears throat> we are still ahead of schedule. <clears throat> We are now talking about the Renewable Energy Directive. Μιλούμε για την οδηγία ανανεώσιμης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το προσχέδιο πράξης κατεξουδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οδηγία για την ε, πρόθεση της χρήσης ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υιοθετήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη. και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Κομισιόν ε, να εκδώσει την ε, κατεξοδότηση πράξη για την ε, χρήση βιοκαυσίμων και για την ε, χρήση της ε, γης, διευρυμένη χρήση γης προς αυτή την κατεύθυνση να σας ενημερώσω ότι έχουμε κρατήσει μία ώρα στο πρόγραμμά μας για αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να παρουσιάσει το προσχέδιο για 15 λεπτά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσίασω αυτήν την έκφραση για ε, τα βιοκαύσιμα υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Η Κομισιόν στις 8 Φεβρουαρίου δημοσίευσε ένα προσχέδιο αυτής της ε, κατεξοδότηση πράξης ε, για μια περίοδο 8 εβδομάδων διαβούλευσης. Για την ακρίβεια 8 εβδομάδων στις οποίες θα πάρουμε το feedback το δικό σας. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να πούμε δύο-τρία πράγματα παραπάνω σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε για το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. το ευρύτερο πλαίσιο αφορά την αναδιατύπωση της οδηγίας ε, για, την, ε, ε για την ενέργεια ως ε, τμήμα του πακέτου που εθετήθηκε πέρσι. Ε, ε, αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ αυτών βιοενέργεια και βιοκαύσιμα. Και ταυτόχρονα το πακέτο αυτό καθορίζει ένα αριθμό σημαντικών απαιτήσεων για το τι είδους βιοκαύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου αυτά να προσμετρώνται στο στόχο. Στους στόχους που θέτει η οδηγία. Επίσης, καθορίζει οι απαιτήσει σε ό,τι αφορά τον, τα βιοκάψιμα υψηλού κινδύνου αλλαγής χρήσης γης και πιο συγκεκριμένα προβλέπει ότι το όριο κάθε κράτους μέλους ε, για τις εκτάσεις που θα ε, θα ε, με προσμετράτε στο στόχο ε, δεν πρέπει να ξεπερνάει το 7% της συνολικής έκτασης. Είναι η προσέγγιση που έχουμε και στην ισχύουσα οδηγία από το 2015. Κάτι που αποτελεί ε, αποτέλεσμα προϊόν τη ισχύουσα νομοθεσία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Στην καινούργια οδηγία που υιοθετήθηκε πέρσι, καθορίζεται ένας στόχος για τα υψηλού κινδύνου βιοκαύσιμα. Ε, η χρήση των βιοκαυσίμων αναφέρεται ότι θα πρέπει να παγώσει κατά την περίοδο 2021-2023 στο επίπεδο που βρίσκεται, που βρίσκεται ε, η η χρήση του το 2019 και μετά το 2023 αυτός ο τύπος βιοκαυσίμων, δηλαδή του υψηλού κινδύνου, θα ε, σταδιακά θα μειωθεί από το 2023 μέχρι το 2030 έτσι ώστε να μηδενιστεί το 2030. Δεν θα είναι πλέον από το 2030 και μετά δυνατό αυτά αυτούς τα βιοκαύσιμα να προσμετρώνται στο στόχο. Επιπλέον υπάρχει εξαίρεση για βιοκαύσιμα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν χαμηλού κινδύνου. Όλα αυτά καθορίζονται σαφώς στην οδηγία Ε, εδώ αυτό το αναφέρει η οδηγία, οπότε δεν είχε και πολλά να κάνει η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τα χαμηλού κινδύνου βιοκάψιμα, η οδηγία αναφέρει ότι μπορούν να παράγονται μόνο από πρόσθετες, ε, εκτροφ, ε, πρόσθετες καλλιέργειες ε, αυξημένης εσοδείας ή από ε, οι οποίες ήδη καλλιεργούνται. Η Κομισιόν απλώ έπρεπε να καθορίσει τα λεπτομερή κριτήρια για αυτή την προσέγγιση και ε, η οδηγία αναφέρει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να βάλει και εκθέσεις ε, για την εξέλιξη της καλλιέργειας ε, φυτών για ανθρώπινη διατροφή και για ζωοτροφές ανακράτος μέλος. Δεν προτείνουμε μια καινούργια πολιτική. Προτείνουμε απλώς τα κριτήρια της προσέγγισης την οποία έχει ήδη συμφωνήσει ο ε, νομοθέτης. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή, τα καλύτερα δυνατά επιστημονικά ε, ε, δεδομένα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας κοινό κέντρο έρευνας. Ε, τα βιοκαύσιμα τα οποία ε, θα ταξινομηθούν σε αυτήν την κατηγορία ε, πρέπει να πληρούν τα εξή κριτήρια. Όλα. Πρώτον, η, η έκταση παραγωγής θα πρέπει να βρίσκεται στο 1% ή 100.000 εκτάρια ετησίως και το 10% αυτών θα πρέπει να βρίσκεται σε γη η οποία να θεωρείται υψηλής αποθήκευσης άνθρακα. Και λαμβάνονται υπόψη και οι εκτάσεις υψηλής απόδοσης. Τώρα, τι σημαίνει σημαντική επέκταση σε γέες υψηλής αποθήκευσης άνθρακα. Ε, αναφέρουμε κριτήρια συγκεκριμένα για να διασφαλιστεί ότι όλα τα βιοκαύσιμα που προσμετρώνται στο στόχο ε, θα οδηγήσουν σε πραγματικές σοβαρές μειώσεις ε, ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αν έχουμε αρνητικές επιπτώσεις όπως απερίμωση ή αποδάσωση, ε, αυτά τα βιοκαύσιμα θα αποκλειστούν. Και βέβαια θα πρέπει να τα συγκρίνουμε με ορυκτούς ε, υδρογονάθρακες, στους οποίους προσπαθούμε βέβαια να αποκαταστήσουμε. Η τα ποσοστά συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα και βασίζονται σε εργασία του Κοινού Κέντρου Έρευνας. Πρόκειται για καύσιμα τον οποίο η, ε, δεν μπορεί να αυξηθεί η συμβολή τους στο στόχο μέχρι το 2023 και από το 2023 και μετά θα πρέπει σταδιακά να μηδενιστούν, να μηδενιστεί η χρήση τους. Δεν μιλούμε για απαγόρευση στη χρήση τους. Ε, απλά από το, 2000, από το 2030 και μετά δεν θα προσμετρώνται στο στόχο τον οποίο έχει θέσει ο νομοθέτης. Τώρα, τα βιοκαύσιμα χαμηλού κινδύνου και εδώ έχουμε ε, ένα αριθμό κριτηρίων. Θα πρέπει να πληρούν τον όρο τα κριτήρια βιωσιμότητας της οδηγίας και μετά έχουμε πρόσθετες ε, καλλιέργειες σε γη η οποία δεν χρησιμοποιείται για τροφή, για παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών ή για ε, γη υψηλής απόδοσης. Αυτά εξαιρούνται από τα κριτήρια υψηλών, υψηλού κινδύνου. Σε... Εκεί έχουμε και κριτήρια συμπληρωματικότητας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο ε, και η πληξιμότητα αυτών των μέτρων θα περιοριστεί στα 10 χρόνια. Μετά έχουμε και απλοποιημένα κριτήρια για πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σχέδια τα οποία χρησιμοποιούν εγκαταλελειμμένη ή ε, υποβαθμισμένη γη, ε, γη η οποία έχει μολυνθεί για παράδειγμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών καθώς επίσης και για μικρές εκμεταλλεύσεις. Αυτά είναι με δύο λόγια τα όσα προτείνει η Κομισιόν. Είναι αρκετά τεχνικά. Το iLook είναι τεχνικό θέμα. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε βρει την πιο ισορροπημένη λύση. Στηριχθήκαμε στα βέλτιστα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία και είμαστε σίγουρα ευθυγραμμισμένοι με, την, με το νομικό κείμενο της ε, για την Ενέργεια. Προφανώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Ε, αν προκύψουν καινούργια στοιχεία. Ε, θα εξακολουθήσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση έτσι κι αλλιώς μέχρι τον Ιούλιο του 2021 θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και, την, ε, και τα επιστημονικά δεδομένα και ενδεχομένως την προσέγγιση μας. Ε, τώρα ε, για τις επόμενες 8 εβδομάδες έχουμε ανοίξει τη διαβούλευση μέχρι τις 8 Μαρτίου. Η Κομισιόν θα διοργανώσει και μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων εκείνη τη μέρα και σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε την κατεξοδότηση πράξη έγκαιρα έτσι ώστε να αυτή να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, πριν την ε, έναρξη της ε, περίοδου διακοπών εργασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Προνώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, παρόλα αυτά είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε. Μετά το Κοινοβούλιο θα έχει δύο μήνες για να εκφέρει αντίρρηση. Σε άλλη περίπτωση ε, δεν θα, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπει σε ισχύ. Περιμένω τα σχόλια των μελών σας. Πρόεδρος, παρακαλώ πολύ ο λόγος στον κύριο εισηγητή, τον κύριο Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα βάλουμε γνώση της πρότασης της Κομισιόν για, την, ε, για τα κριτήρια τα οποία θα καθορίζουν τα βιοκαύσιμα υψηλού και χαμηλού κινδύνου ε, ε, αλλαγής χρήσης γης. Όλοι μας γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της οδηγίας ανανεώσιμων ενέργειας. Τελικά καταλήξαμε νομίζω σε μια λογική σε ένα λογικό συμβιβασμό. Ε, είναι μια σημαντική πρόκληση το να βρούμε λύσεις ε, για να ε, περιορίσουμε την αλλαγή χρήσης γης προκειμένου να παραχθούν βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς διότι αυτά τα βιοκαύσιμα δημιουργούν προβλήματα και στην απασχόληση και, στη, και προβλήματα αποδάσωσης ε, και προβλήματα εκπομπών. Η οδηγία εντοπίζει ποιες είναι, ποια είναι τα βιοκαύσιμα υψηλού κινδύνου και ποια είναι χαμηλού κινδύνου, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο. Όπως και στην οδηγία, επιτρέπει, επιτρέπει έτσι ε, να τη χρήση ε, βιοκαυσίμων ε, στην περίπτωση που αυτά είναι χαμηλής, χαμηλού κινδύνου, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Παρ' όλα αυτά, από όταν δημοσιεύθηκε το προσχέδιο αυτής της κατεξιδότησης πράκτης, ε, πολλές ε, φωνές ισχυρίζονται ότι αν θέλουμε να λύσουμε μια και έξω αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να κλείσουμε, να καλύψουμε τα κενά, τα παραθυράκια τα οποία υπάρχουν, να κλείσουμε τις πίσω πόρτες ε, οι οποίες ε, ως κερκόπορτες θα μπορούσαν να καταστρέψουν όλο το οικοδόμημα αυτής της ε, βιώσιμης παραγωγής βιοκαυσίμων. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, δεν υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα για το όριο του 10%. Ε, γεών με υψηλή αποθήκευση άνθρακα. Είναι χαμηλότερο από το 14% στο οποίο γίνεται αναφορά στην έκθεση. Για ποιο λόγο προτείνεται 10% και όχι ε, κάτι ε, ακόμα χαμηλότερο και προφανώς πιο περιβαλλοντικά φιλικό προς το περιβάλλον. Δεύτερον, καθορίζονται τα κριτήρια Προσθετικότητα, συμπληρωματικότητα για την αδειοδότηση, για την ε, πιστοποίηση. Αλλά κάποιε οργανώσει αναφέρουν ότι υπάρχουν κενά τα οποία θα επιτρέψουν να πάρουν πιστοποίηση ω χαμηλού κινδύνου βιοκαύσιμα, τα οποία δεν είναι χαμηλού κινδύνου. Για παράδειγμα, μικρές εκτάσεις, ε, μικρότερες των 2 ή των 5 εκταρίων ή εγκαταλειμμένες Yes. Ε, μετρήσατε τον αντίκτυπο αυτού του μέτρου, αυτού του όρου. Έχουμε την ευκαιρία να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα βιοενέργειας, ε, αποδάσωσης και εκπομπών. Χρειαζόμαστε όμως καθαρούς κανόνες, σαφή και βάσιμα κριτήρια και επαρκή έλεγχο. Για να στηρίξουμε αυτή την κατεξοδότηση πράξη, η Κομισιόν θα πρέπει να αναθεωρήσει την πρότασή της. Η βιώσιμη βιοενέργεια είναι απολύτως απαραίτητη για να επιτύχουμε την ουδετερότητα εκπομπών ε, και προκειμένου ο κόσμος να γίνει βιώσιμος. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Κέλλη του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Κομισιόν για τις εξηγήσεις που έδωσε για την εκτελεστική πράξη. Λογικά πράγματα είπατε και βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα. Όμως, όπως λέει ο κ. Μπλάνκο, υπάρχουν και ερωτήσεις. συμφωνούμε ότι πρέπει να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση εκπομπών οξυδίων του άνθρακος και από τα βιολογικά καύσιμα. Ερωτήσεις. Πρώτη. Αν το Κοινοβούλιο προβάλλει ένσταση, και μάλλον θα το κάνει, φτάνεται πια Μάιο-Ιούνιο. Άρα προχωρείτε στο επόμενο Κοινοβούλιο για να μπορέσει να τελικοποιηθεί η πράξη. Δεύτερο, ο κύριος Λόπες μίλησε για το 10% αλλά αυτό μου φαίνεται αυθαίρετο. Εκεί μπορεί να μπει και η σόγια ενδεχομένω. Αυτό σκέπτεστε. Γιατί αυτά τα συζήτησε ο πρόεδρος Γιούνκερ με τον πρόεδρο Τραμπ. Και για τις μη χρησιμοποιούμενες και εγκαταλελειμμένες γέες. Πώς εκτιμάτε τις συνέπειες αυτών, μάλλον στις γέες αυτές. Και η, ποια, ποια θα είναι η επίπτωση αν επεκταθεί και σε μη χρησιμοποιούμενες γέες. Αυτά όλα θα πρέπει να συμμορφώνονται και με τους κανόνες του ΠΟΕ, υποθέτω. Και το 10% θα συμπορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ και θα είναι αποδεκτό από αυτόν. Τέλος, πώς θα τα παρακολουθείτε όλα αυτά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσετε ότι ό,τι προτείνετε τελικώς θα εφαρμόζεται. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ θα έπρεπε να λάβω τον λόγο, αλλά ο κύριος Κέλλη έκανε ήδη τις ερωτήσεις που θα έκανα και εγώ. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Μέτς των Πρασίνων. Συγγνώμη, πρόκειται για την κυρία Μέτς. Η κυρία Μέτς, κύριε Πρόεδρε, μην ανησυχείτε όμως, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν, για την παρουσίαση. Οφείλω να σας μεταφέρω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η πρότασή σας δεν έρετε στο ύψος των τρέχουσων προκλήσεων. Προσπαθείτε ε, να παίξετε τον εξισορροπητή ανάμεσα στην εμπορική πολιτική και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όμως δεν μπορείτε να τα περιλάβετε όλα και προτείνετε τελικά ένα κείμενο το οποίο εξασφαλίζει το status quo, το είπατε και στους ίδιους. Δηλαδή την ε, μαζική χρήση βιολογικού καυσίμου στη βάση φινικελαίου στην Ευρώπη. Έτσι δυστυχώ, οι πράξεις, προτείνετε, οι πράξει σα μάλλον δεν συμβαδίζουν με τα λόγια σα. Αφενό αναγνωρίζετε τις καταστροφικές συνέπειες ε, των φυτιών ε, φινικελαίου για το κλίμα, για τη βιοπικιλία και για τα δικαιώματα των ντόπιων πληθυσμών. Από την άλλη μεριά δυστυχώς ανοίγετε πόρτες και παράθυρα σε υπέρμετρες χρήσεις που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να συνεχίσει να εισάγει τεράστιες ποσότητες φινικελαίου που έχει παραχθεί με μη βιώσιμο τρόπο. Διότι πρώτον, τίποτε δεν επιτρέπει να πει κανεί ότι οι εκμεταλλεύσει μικρού μεγέθου είναι πιο ενάρετε από τι μεγάλε σε ό,τι αφορά ε, τις περιβαλλοντικές συνέπειες και όλοι γνωρίζουμε την δημιουργικότητα των πολυεθνικών για να κατακαιρματίζουν ε, τις εκμεταλλεύσεις, να ε, ανακατεύουν τους τίτλους ιδιοκτησίας και να προστατεύονται έτσι. Από την άλλη μεριά, ε, ο όρος μη χρησιμοποιούμενες γέες, που δεν είναι και απόλυτα κατάλληλος, διότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι γης είναι χρήσιμες για τη διατήρηση της βιοπικιλίας και για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Τρίτο, είναι απόλυτη ψευδέστηση να περιμένετε από διαδικασίες πιστοποίησης να είναι αξιόπιστες, ενώ συχνά καταλήγουν να είναι ένα είδος greenwashing σε μεγάλη κλίμακα. Τέλος, το συμπέρασμα είναι ότι ενώ παρουσιάζεται τις σχέσεις μας, τις εμπορικές σχέσεις με Ινδονησία και Μαλαισία, αποφασίζετε εσείς να θυσιάσετε το τροπικό δάσος και με τον ίδιο αυτό εμπορικό ρεαλισμό που σας οδηγεί να μην αντιμετωπίσετε το ζήτημα της σόγιας ενώ η σόγια είναι βιολογικό καύσιμο το οποίο αποδίδει στην ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερες εκπομπές οξυδιών του ανθρακός. Τελικώς αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι οι μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες εκμεταλλεύονται το φινικέλαιο και την σόγια περιφρονώντας τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κανόνες. Και ως συνήθως το κλίμα, η φύση, τα ζώα και τέλος η ίδια η ανθρωπότητα είναι τα μεγάλα θύματα. Κύριε, Προ... Επίτροπε, μάλλον δεν είναι πέραν ο Επίτροπο, αλλά αυτό μεταφέρεται το μήνυμα. Ελπίζω η Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγισή της και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία πρόταση εφαρμοστικής πράξης που να μην σημαίνει στασιμότητα, αλλά πραγματικά προοδευτική. Να είναι πραγματικά προοδευτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαρτάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μέση με κάλυψε εν μέρη. Βεβαίως πάντα είναι καλό να μπορεί να επαναλαμβάνει κανεί σωστά επιχείρηματα. Όταν άκουσα για την εκτελεστική πράξη της Κομισιόν, ανεφώνησα και είπα εδώ μας λένε τρελά πράγματα. Η ερώτηση που προέκυψε είναι ποια ανταλλάγματα δίνουν Μαλέοι και Ινδονήσιοι για να προτείνετε αυτό που προτείνετε. Διότι μιλείτε πολύ για επιστημονικά ε, δεδομένα, τα οποία ούτω ή άλλω είναι αμφισβητούμενα, Ποτέ δεν μιλήσατε όμως για κοινωνικά δεδομένα. Γνωρίζετε ότι κάθε Πέμπτη μαζεύονται εδώ χιλιάδες νεαρών διαδηλωτριών και διαδηλωτών που μας λένε σταματήστε επιτέλους την σφαγή. Η απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις σημαντικές ευρωεκλογέ είναι «Μα μη σας νοιάζει, προχωρήστε, δεν υπάρχει τίποτα να δείτε εδώ». Και είναι πολύ πιο σημαντικό το διεθνές εμπόριο από το μέλλον του πλανήτη. Μήπως έχουμε τρελαθεί τελείως. Και τέλος είναι και πολύ άσχημο το μήνυμα που δίνεται, διότι όπως είπε πριν η κυρία Μέτς, δίνεται εμπιστοσύνη στις πολυεθνικές ώστε να φροντίσουν αυτές ότι θα είναι μικρές οι εκμεταλλεύσεις για να μπαίνουν στα κριτήρια εξαιρέσεων που υποβάλλεται. Γνωρίζετε πολλές μη χρησιμοποιούμενες γέες σε αυτές τις περιοχές του κόσμου όπου οι διατροφικές ανάγκες αυξάνονται διαρκώς και μάλιστα σε βάρος του, της ε, βιοπικιλότητας και της ισορροπίας. Απορρίπτω την πρόταση και ελπίζω η διαβούλευση που θα οργανώσετε με την κοινωνία των πολιτών θα σας δώσει ένα ηχηρό όχι, το ελπίζω, διότι ήδη το βιολογικό καύσιμο που προέρχεται από ε, φινικέλαιο είναι μια αντίφαση. Η ίδια η Κομισιόν λέει ότι το φινικέλαιο είναι το πιο ε, βλαβερό καύσιμο. Δεν το λέτε εσεί προσωπικά, το λέει η Κομισιόν. Και να όμω που προβλέπετε την εξαίρεση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι τα ανταλλάγματα που θέτουν επιτάπητο Μαλαισία και Ινδονησία για να ανοίξει τι εξαιρέσει αυτέ τι οποίε εξηγήσατε. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις, δεν φαίνεται. Οπότε ο κύριος Βανστίν θα πρέπει να δώσει τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα τις μεταφέρω στον Επίτροπο που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Αλλά ας προσπαθήσω να δώσω κάποιες εξηγήσει γύρω από τα θέματα τα οποία θέσατε τα, με ιδιαίτερα έγκριτο τρόπο. Για τον κύριο Μπλάνκο Λόμπες, σχετικά με τα ανώτατα δεν είναι μεταξύ μας πια. Αλλά το 10% και ο λόγος για τον οποίο εξελέγει, εμείς ε, αποδεχθήκαμε ένα αρκετά συντηρητικό ποσοστό για να διασφαλίσουμε ε, ότι δεν είναι σημαντικές οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σαφές επίσης ότι μέσω του συγκεκριμένου ορίου, και έρχομαι εδώ και στις υπόλοιπες παρατηρήσεις, ότι το φινικέλαιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των βιοκαυσίμων υψηλού κινδύνου και δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο ε, εσείς λέτε ότι εγκρίνουμε και παρατείνουμε το status quo ίσα ίσα διευρύνουμε τις ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε τα βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται ε, να παρουσιάσουν εκ σημαντικές μορφές εξοικονόμησης στον τομέα των εκπομπών, να μην οδηγούν σε αποψήλωση των δασών και να μην απορροφούν αρρώσιμες γέες. Συνεπώς λοιπόν η χρήση των βιοκαυσίμων και του φινικελαίου ως βιοκαυσίμου ε, θα καταργηθεί εκτός από ορισμένες ακραίες περιπτώσεις όπου ε, επιβεβαιούται ο χαμηλός κίνδυνος. Οι περιπτώσεις αυτές, οι εξαιρέσεις αυτές θα είναι καθορισμένες με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο και μόνο όταν είναι προφανές ότι ε, υπάρχει προσθετικότητα με τις υπόλοιπες καλλιέργειες και ότι υπάρχουν μικροί παραγωγοί οι οποίοι ε, θα δυσκολευθούν ιδιαίτερως να περάσουν σε αλλαγή καλλιέργειας και είναι απαραίτητο αυτό για τις πρακτικές τους. Τώρα για το 10% εμείς θεωρούμε ότι είναι το σωστό ποσοστό. Είναι πιο αυστηρό από το 14% το οποίο προτείνεται σε άλλα σημεία. Και αποκλείει η Φινικέλεα τα οποία ε, έχουν ε, ε, συνεισφέρει ιδιαιτέρως στην κατάκτηση σε εισαγωγικά νέων γεών για καλλιέργεια στο παρελθόν. Εμείς τώρα για τους ε, μικρούς καλλιεργητές το έχουμε βάλει σε εισαγωγικά, είχαμε κάνει αρκετές συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα και θα θέλαμε να δούμε τι αντιδράσεις υπάρχουν. Είπαμε ανάμεσα στο 2 με 5 να μείνουμε και φυσικά θα θέλαμε να δούμε και τα επιχειρήματα ε, σχετικά με τον ορισμό του μικρού καλλιεργητή. Τώρα τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις από τον κύριο Κέλλη και για τη σόγια. Πιστεύουμε ότι η σόγια είναι διαφορετικό πράγμα από το φινικέλαιο. Αν δείτε τους αριθμούς θα δείτε ότι δεν υπάρχει τέτοια διεύρυνση των καλλιεργειών ε, σε αρρώσιμες γέες από την σόγια όπως από το φινικέλαιο τα βιοκαύσιμα από τη σόγια μπορούν να παρουσιάζουν πιστεύουμε εξοικονομήσεις εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει όμως πάντα η δυνατότητα της αλλαγής αυτών των χαρακτηριστικών και γι' αυτό εμείς παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά τις πιθανές αλλαγές και αν χρειαστεί θα αλλάξουμε την ε, θέση μας και τις ρυθμίσεις όπως προβλέπεται στα παρατήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή είναι απολύτως συμβατή με τον ΠΟΕ. Ε, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Δεν ε, ξεχωρίζεται ένα κάποιο βιοκαύσιμο ή βάρος κάποιο άλλο. Εμείς απλά χρησιμοποιούμε το κριτήριο του χρήσιμου βιοκαυσίμου μέσω αυτών των αντικειμενικών κριτηρίων βλέπουμε ποια είναι τα καύσιμα που παρουσιάζουν υψηλούς ή όχι κινδύνους. Είμαστε σε θέση να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά πολύ καλύτερα από το, το παρελθόν, μέσω ακριβώς και εικόνων δορυφορικών, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιώντας και άλλα κριτήρια αηφορίας, μπορούμε να επιβάλλουμε ε, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της κατάστασης. Νομίζω ότι απάντησα στην ερώτηση της κυρίας Σμέτς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε τις ποσότητες με ξεκάθαρο αξιόπιστο τρόπο και νομίζω ότι οι πιστοποιήσεις είναι αυτές οι οποίες χαρακτηρίζουν και τους κανόνες αηφορίας. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τα κριτήρια αυτά αηφορίας για τον χαρακτηρισμό των βιοκαυσίμων. Για τη σόγια νομίζω ότι έδωσα ήδη απάντηση. Δεν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι το ίδιο με ότι με το φιλικέλαιο, με το φινικέλαιο. Άκουσα ότι εσείς αποφασίσατε ότι θα απορρίψετε την κατεξουσιοδότηση πράξη, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια νέα πρόταση στα πλαίσια της επόμενης κοινοβουλευτικής περίοδου βέβαια, γιατί ε, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει σύντομα. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες από τις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε. Βρισκόμαστε τώρα στην διαδικασία διαβούλευσης. Έχουμε προσκαλέσει εμπειρογνώμονες από όλη την γάμα θα έλεγα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Φυσικά και οι εκπρόσωποι και οι εκπρόσωποι εννοώ και οι εμπειρογνώμονες στους οποίους θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει μπορούν να εμπλακούν με κάποιο τρόπο. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Αλλά όπως είπα στην αρχή αυτή την ξεκάθαρη απόφαση την οποία πήραν οι συνομοθέτες μέσω της βασικής οδηγίας. Καθορίζεται η πολιτική, γενικά βέβαια μπορεί κανείς να πει ότι οι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι ρυθμίσεις οι οποίες ε, προτείνονται μας ε, επιτρέπουν να κρίνουμε τα προϊόντα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου και έτσι να ανταμείψουμε και τους παραγωγούς οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν το προσθετικό στον τρόπο παραγωγή τους και να αποδείξουν ότι δεν διευρύνουν τις καλλιέργειές τους σε υψηλών εκπομπών εκτατικές καλλιέργειες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και το Κοινοβούλιο τελικά θα υποστηρίξει την πρότασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας από εδώ και πέρα για οποιαδήποτε μορφή διμερούς επικοινωνίας, για τεχνικές λεπτομέρειες. Μπορείτε να συζητήσετε και με τους εμπειρογνώμονές μας για όλα τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Βανστέν. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και για τις ερωτήσεις σας. Εμείς είμαστε αρκετά νωρίς στο πρόγραμμά μας. Περνάω στο επόμενο θέμα. Είναι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις εν εξελίξη. Θα μιλήσουμε και για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση του προγράμματος πλαισίου έρευνας Horizon Europe. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καθορίζει τους τρόπους συμμετοχής και διάδοσης των ρυθμίσεων που περιλέχει. Να υπενθυμίσω ότι ο δεύτερος τριμερής διάλογος έγινε την 29η Ιανουαρίου και θα ήθελα αμέσω να δώσω το λόγο στον κύριο Ντανίκα για δύο λεπτά. Καλό σας απόγευμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχει καμία μείζον εξέλιξη από την τελευταία ενημέρωση που σας έκανα. Σήμερα διεξήχθη συνάντηση του Συμβουλίου και περιμένουμε ακόμη να δούμε ποια θέση θα διαμορφώσουν διότι μέχρι τώρα η θέση τους δεν ήταν ιδιαίτερα εύκαμπτη διάλογος θα γίνει την Πέμπτη, ώστε όλα τα σημαντικότερα θέματα θα συζητηθούν εκεί, την Πέμπτη. Και θα σας ενημερώσουμε. Δυστυχώς για την ώρα, μηδέν πρόοδος σε όλα τα μείζωνα θέματα, η ΑΕΣΥ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαδικασίες fast track, διεύρυνση και ούτω καθεξής πολύ σύντομη όπως ακούσατε ενημέρωση από τους δύο πρώτους τριμερείς διαλόγους. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Φαίνεται πως είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Ο επόμενος τριμερής διάλογος, όπως εξηγήσατε, είναι την 5η, δηλαδή 21 Φεβρουαρίου, 21 Φεβρουαρίου, έτσι είναι. Α, με συγχωρείτε, κυρία Τόγια, δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο είπα και στον συνάδελφο Νίκα επανειλημμένα, ότι κατανοώ την δυσκολία που παρουσιάζει το θέμα αυτό, ένα περίπλοκο θέμα όπως είπατε, τεχνικά δύσκολο και παρακολούθησα γενικά τον τρόπο με τον οποίο προώθησε το θέμα ο συνάδελφος εισηγητής ora o come un punto eh, noi, lui Νομίζω ότι η πρωτοβουλία η οποία είχε προβλεφθεί σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μια ad hoc πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει στο σύνολο των μικρομεσαίων και να έχει σαν στόχο την αύξηση της δραστηριότητάς τους, και μάλιστα είχαν προβλεφθεί από πλευράς μας δύο δις επιπλέον, θα ήθελα να μάθω σε ποιο τρόπο ε, το μέτρο αυτό έχει προχωρήσει. Τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία, σαν παράδειγμα. Έχει αλλάξει κάπως ε, η αρχική ρύθμιση. Μήπως θα μπορούσαμε εμείς μέσα σε αυτά τα δύο δις τα οποία έχουμε προαποφασίσει κάποια πιο συγκεκριμένα μέτρα διότι αλλιώς θα πρέπει να καθορίσουμε κάποια συγκεκριμένα ποσοστά. Να πούμε ας πούμε ότι το 75% θα πάει σε μικρομεσαίες είτε στο δεύτερο πυλώνα είτε στο τρίτο πυλώνα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας καθορισμένος κύκλος μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να αποδείξουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σαν μικρομεσές, τις μικρομεσαίες δεν τις εγκαταλείπουμε και ότι για μας παραμένουν σημαντικές για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι βασικό, είναι καθοριστικό για μας, γιατί αλλιώς λέμε ότι είμαστε η φωνή των μικρομεσαίων, αλλά δεν το κάνουμε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο και σε επίπεδο Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Συμβουλίου. Πάντως, έχει υπάρξει ήδη μια απόφαση του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που είναι μεταξύ μας και ο συνάδελφος Έλα, γιατί ξέρει και αυτός ποια είναι η απόφαση την οποία έχει πάρει το Κοινοβούλιο, ακόμα και αν αλλάζει κάπως προϋπολογισμό, ε, συγγνώμη, προσανατολισμό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Κύριε Νίκα, θέλετε να απαντήσετε. Να επιβεβαιώσω ότι το θέμα αυτό είναι πάντα υποσυζήτηση. Τώρα τα 2,5 δις λέει ο κύριος Νίκα. Δεν έχουν συζητηθεί ακόμα στο Συμβούλιο. Ήταν τμήμα της δικής μας πρότασης και το 70% οριζόντια κατανομή για τις μικρομεσαίες και αυτό είναι κάτι που δεν έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο. Υπάρχουν δύο επιλογές εδώ. Αν το Συμβούλιο επιδείξει την ευελιξία που χρειάζεται στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, τότε θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μέσα σε ένα μήνα, το Μάρτιο. Αν όχι, το Κοινοβούλιο θα κλείσει τις διαπραγματεύσεις το Μάρτιο μεν του 20 δε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς έχουμε μια σαφή εντολή από πλευράς μας, σχεδόν ομοφωνία από όλες τις πολιτικές ομάδες και στο Συμβούλιο έχουν κάποιες θέσεις ε, χωρίς καθόλου ευελιξία και δεν δίνουν ξεκάθαρη εντολή να διαπραγματευτούν ούτε καν το 1%. Συνεπώς είναι αδύνατο να αλλάξει η κατάσταση έτσι. Λοιπόν, ή θα πρέπει να διαπραγματευτούν και να κάνουν συμβιβασμούς ή το επόμενο κοινοβούλιο, τον Μάρτιο του 20, θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις αυτές. Πράγματι είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα αυτό. Ο κύριος Έλα έχει το λόγο. Πράγματι είναι περίπλοκο από τη μία οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν τα πιο σημαντικά τα θέματα και από την άλλη δεν θα πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ γιατί ίσως δεν χρειαστεί να υποχωρήσουμε τελικά. Το η σοσιαλιστική ομάδα σαν παράδειγμα επιμένει σε σχέση με τα ειδικότερα προγράμματα για τις μικρομεσαίες. Εμείς σαν ΕΛΚ θέλουμε να δούμε κάποιες μικρές βελτιώσεις σε σχέση με το λεγόμενο fast track είναι λοιπόν σαφές ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες το Κοινοβούλιο δεν θα εγκαταλείψει κάποιες από τις βασικές του θέσεις. Τώρα, είναι καλό να γίνει η διαπραγμάτευση στο επόμενο Κοινοβούλιο στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και γίνουν δεκτές οι θέσεις των πολιτικών ομάδων, ε, νομίζω ότι θα διαπραγματευτούμε τον προϋπολογισμό με πολύ μεγαλύτερη άνεση. Στο παρελθόν είχαμε δεδομένη την κάλυψη, την δημοσιονομική, την προϋπολογιστική και μπορούσαμε να εκλεπτύνουμε στην πρότασή μας. Αν υπάρξει λοιπόν επί τη βάση της αρχής μια συμφωνία με το Συμβούλιο, τότε θα είμαστε πραγματικά σε πιο καλή θέση για να διαπραγματευτούμε και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, για το Συμβούλιο να ε, ζητήσει να γίνουν μειώσεις στον προϋπολογισμό. Σε επίπεδο τακτικής δηλαδή πρέπει να επιμείνουμε για μία εκ των προτέρων συμφωνία. Γνωρίζοντας ότι για τον προϋπολογισμό τα συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία θα τα θέσουμε σε συζήτηση τον επόμενο χρόνο. Πάντως, σε επίπεδο αρχής, καλό είναι να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία τώρα, πρακτικά τώρα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της νομικής βάσης, αναφερόμεθα σε μια λύση η οποία θα είναι ιδιαίτερος περίπλοκη. Θα δημιουργηθούν συνθήκες τριμερούς διαλόγου που θα βασίζεται στη συμφωνία για την καλύτερη διαπραγμάτευση και ε, την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε πάντως εξελίξει τον τριμερή διάλογο και γι' αυτό θα πρέπει οι συμβιβαστικές λύσεις τις οποίες θα καταλήξουμε να είναι λειτουργικές και θα ελέγξουμε αν, είναι, αν σέβονται και αν είναι σεβαστές, ε, συμβατές με, ε, την, ε, με τις πολιτικές μας αποφάσεις. Αλλιώς τα πράγματα θα μείνουν στάσιμα. Έχουμε πολλά θέματα στο pipeline πολλά από τα θέματα αυτά έχουν τύχει μιας κάποιας χρηματοδότησης. Το πρόβλημα είναι στην παρούσα φάση ότι λόγω της περιπλοκότητας των θεμάτων αυτών υπάρχει καθυστέρηση. Και δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε σε, στον καθορισμό λεπτομεριών εφαρμοστικών Έχουμε κάποια στοιχεία για το Horizon Europe. Αλλά το 2020 δεν θα έχουμε να κάνουμε με το Horizon 2020, αλλά το τι θα περιλαμβάνεται στο επόμενο δημοσιονομικό. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ε, ποιοι είναι οι βασικοί μας στόχοι όπως το κάνουμε τώρα σε σχέση με το Horizon 2020. Μήπως θα πρέπει να τους κάνουμε να περιμένουν πριν καταλήξουμε στις τελικές μας αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει το 2021. Αλλά τότε δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την προπαρασκευαστική θάση. Συνεπώς όλα αυτά δείχνουν ότι σε επίπεδο τακτικής θα έπρεπε να προχωρήσουμε γρήγορα. Ήδη με το Brexit βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τα επόμενα προγράμματα upfront εκ των προτέρων και αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση. Πρέπει να περάσουμε σε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις εγώ θέλω να αποφύγουμε ε, τις κατά πλειοψηφία θέλουμε ομοφωνίες γύρω από το θέμα αυτό. Αν δεν δουλέψει θα δούμε τι να κάνουμε. Αν δουλέψει όμως τότε θα έχουμε κάνει πολλά για τους μικρομεσαίους, για τους πολίτες της Ένωσης και θα βρεθούμε σε ισχυρότερη θέση και στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις το 20. Οπότε τότε το Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το τι θέλει να διώξει και τι θέλει να κρατήσει. Πρέπει λοιπόν να φανούμε φιλόδοξοι. Πρόεδρος, καλά λοιπόν. Είναι πράγματι περίπλοκο το θέμα. Θα προχωρήσω όμως στο επόμενο τώρα. Το ίδιο περίπλοκο. Τόσο πολύ μάλιστα που χρειάστηκε να αναβληθεί. Άρα, εκφωνώ τώρα το επόμενο θέμα, το επαριθμό 15, θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021 έως 27. Και ο πρώτος τριμερής διάλογος έλαβε ήδη χώρα στις 13 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε εκεί και μάλιστα δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Μλινάρ είναι λίγο πιο απλό το θέμα αυτό και με πολύ θετική έκβαση. Όπως είπατε πολύ σωστά την περασμένη Τετάρτη ολοκληρώσαμε επιτυχώς το, τη μοναδική, πρώτη και μοναδική συνάντηση του τριμερούς διαλόγου. Το Συμβούλιο ήταν πολύ επικοδομητικό, έδειξε πνεύμα συνεργασία. Αυτό μας επέτρεψε να καταλήξουμε στη συμφωνία στα εκρεμή πολιτικά θέματα μετά από έξι γύρους τεχνικών συναντήσεων. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι ισορροπημένο διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και τους στόχους του μεταξύ των πολιτικών θεμάτων που διαπραγματευτήκαμε, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής. Πρώτον, η εφαρμογή των στόχων διευκρινίστηκε έτσι ώστε ο αυτός κανονισμός να ενταχθεί στο υπάρχον πλαίσιο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα. Μόνο μέσω συνεργειών μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν διατηρεί ένα περιθώριο ελιγμών έτσι ώστε να διαχειριστεί το πρόγραμμα μέσω της άμεσης εφαρμογής. Δεύτερον, εξασφαλίσαμε ε, ισχυρό σεβασμό της ιδεοντολογικής διάστασης, ιδιαίτερα για το στόχο 2 της ε, τεχνητής νοημοσύνης, ε, υπόψη τις κατευθύνσεις γραμμές τις οποίες ε, θα καθορίσει η ομάδα ad hoc για την ε, τεχνητή νομοσύνη η οποία θα ε, ε, συστήσει η Κομισιόν. Αυτή, με βάση αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές θα γίνεται έλεγχος για τη συμμόρφωση των υποβαλλόμενων προσχεδίων. Επίση, ε, τη συμφωνία για τα ευρωπαϊκά hubs καινοτομία, ψηφιακή καινοτομία, ε, προκειμένου η διαδικασία να είναι ε, συναγωνιστική, ανταγωνιστική. Υπάρχουν βέβαια κάποια οριζόντια θέματα τα οποία έχουν σχέση με το πολιτές πλαίσιο, τα οποία δεν συζητήσαμε, αλλά καταλήξαμε σε όλα τα υπόλοιπα. Διατηρούμε βέβαια την ε, θέση μας όπως την ψηφίσαμε το Δεκέμβρη στην Ολομέλεια για τα θέματα που δεν ήταν ανοιχτά προ διαπραγμάτευση, 7 ακριβώ τα οριζόντια θέματα που αφορούν συνολικά το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Περιμένουμε και την γραπτή επιβεβαίωση του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν που βοήθησε πάρα πολύ καθ' όλη τη διαδικασία, καθώς επίσης και την Ρουμανική Προεδρία για τις ε, γενναίες προσπάθειες που έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή των διαπραγματεύσεων. Και βέβαια ο κύριος Μπούζεκ δεν είναι εδώ, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, ο οποίος προείδευσε του τριμερούς διαλόγου. Τέλος, να ευχαριστήσω την γραμματεία και το προσωπικό αυτής. Ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστούμε για τα χειροκροτήματα, κυρίως για τον κύριο Μπούζεκ και για το προσωπικό. Παρακαλώ πολύ, ενημερώστε τον κύριο Μπούζεκ για τους επένους οι οποίοι ακούστηκαν και τους οποίους σίγουρα αξίζει. Περάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Ο τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 22 ε, Ιανουαρίου. Μια, μια επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα σήμερα σήμερα το βράδυ. Ο λόγος στην κυρία Βερκούνεν, Βίρκουνεν να μας ενημερώσει για τον, την πρώτη συνεδρία του τριμέρου διάλογου. Ναι, ήδη σας είχα ενημερώσει ε, για το τι θα συζητούσαμε. Ε, εστιάσαμε στο τμήμα των μεταφορών στην τελευταία μας συνεδρίαση. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τις μεταφορές. Δεν ακουμπήσαμε και πολύ θέματα ψηφιακά ή ενέργειας. Συνεδριάσεις είναι τεχνικής φύσεως, ε, ε, μάλλον έχουν γίνει και τεχνικής ε, φύσεως συνεδριάσεις, έχουν προχωρήσει. Μετά τη σημερινή θα έχουμε άλλη μία συνάντηση του τριμερούς διαλόγου και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουμε τελικά το Μάρτιο, έτσι ώστε στην κοινή συνεδρίαση επιτροπής με την ΤΡΑΝ να ψηφίσουμε και να, το θέμα να περάσει στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Πάντως δεν συζητήσαμε ψηφιακά θέματα και θέματα ενέργεια του Σοπολίω ως τώρα. Ίσως να ξεκινήσουμε σήμερα το βράδυ. Αν δεν επέλθει συμφωνία λοιπόν σήμερα το βράδυ, ήδη έχετε προγραμματίσει στις 7 Μαρτίου επόμενη συνάντηση. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί αυτή η τελευταία συνάντηση να λάβει χώρα. Στα διάφορα υπάρχει κάτι? Όχι. Ωραία. Να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για τις 4 Μαρτίου έχει ακυρωθεί ακυρώθηκε. Οπότε η επόμενη συνάντηση θα, συμβεί, θα λάβει χώρα πραγματικά στις 18 Μαρτίου Δευτέρα από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Κλείνω τη συνεδρίαση και ευχαριστώ τους πάντες για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστώ.